Guten Morgen. Ich hoffe, wir können anfangen. Ich mir diese Präsenz auch Καλημέρα σα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε τόσο πολύ άριθμοι. Ε, θα είχα χαρεί πάρα πολύ αν είχατε έρθει και χτε και θα είχατε βγει κερδισμένοι, γιατί χτε είχαμε μια θαυμάσια ακρόαση με θέμα την δημιουργική Ευρώπη. Χάσατε πάρα πολλά. Ειλικρινά, ήταν μια από τι καλύτερε ακροάσει που είχαμε τον τελευταίο καιρό. Λυπάμαι που δεν ήρθατε. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Πάμε στο σημείο υπαριθμών 7. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Φλωρεντίας. Νομίζω μιλήσαμε χτες ε, γι' αυτό και η ψηφοφορία είναι μόνο με ναι ή όχι. Και όπως σας είπα και χθες, εντωμεταξύ άξιζε τον κόπο που κοιτάξαμε λίγο το όλο θέμα, διότι το κείμενο που είχε προτιμάσει η Κομισιόν δεν ήταν καλό. Δεν είχε ετοιμάσει, δεν είχε προσφέρει σχεδόν τίποτα. Ούτε το Συμβούλιο το είχε δει το κείμενο. Εμείς ε, το εξετάσαμε, αλλάξαμε ό,τι μπορούσε να αλλάξει. Ε, κατόπιν του του ε, ήταν πολύ καλή αυτή η δουλειά και σας παρακαλώ να ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Πρέπει να ψηφίσουμε με ε, την κάρτα μας ηλεκτρονικά. Ε, άρχισε η ψηφοφορία. Έκλεισε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην ε, επόμενη ψηφοφορία, Νάντια Χίρς, πρόκειται για μία μελέτη σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα. Κυρία Χίρς, θέλετε να πείτε κάτι? Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να ευχαριστήσω θερμά για την πολύ καλή συνεργασία ε, με τους σκιώδεις εισηγητές. Ξέρω πολύ καλά ότι στην ε, γνωμοδότηση προέκυψαν πολλές τεχνικές ε, δυσκολίες. Ξέρετε πώ είναι το πρόβλημα όταν είναι κανεί παράλληλα σε δύο επιτροπές. Ε, νομίζω όμως ότι είναι πάρα πολύ καλή έκθεση και γι' αυτό υπερψηφίζω. Πολύ ωραία. Πάμε στην ε, τροπολογία υπερθμών 17. Ποιος είναι παρακαλώ υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. 12 με 9. Λοιπόν, 12 με 10 εγκρίνεται. Πάμε στο 18, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. 19, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το 20, υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το 24 ε, καταπίπτει. Πάμε στο 25 υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται. Το 26 υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται, το 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 28 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίδων. The vote is closed. Έκλεισε η ψηφοφορία. 10 με 11 απορρίπτεται. Γεια. Sì, non io. so. Come Lei ha votato come? Contro. Yeah, yeah, ja. Contro. So, mi va? Abbastanza. Contro. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται όχι μισό λεπτό, 43 παρακαλώ, υπέρ κατά, αποχές ε, εγκρίνεται, 44 υπέρ κατά, αποχές ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για το 44. Έκλεισε. Ο κύριος Πιτέλα. Υπέρ. Απορρίπτεται. 7 προς 16, 17 λέει πρόεδρος, ε, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. 13 εγκρίνεται. 48 υπέρ. Εγκρίνεται. Α, ε, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Το 50 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Αρχίζει η ψηφορία. The vote is closed. 11 12 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται. Το 1 υπέρ, κατά, αποχές ε, ηλεκτρονικός έλεγχο. The vote is closed. 13 against. 13 zu 12 angenommen. Which one? Uh, Εγκρίνεται. Äh, Amendment 2. Τροπολογία 2. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Το 8. Έκλεισε η ψηφοφορία. 14 με 11 εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ κατά αποχές σε ηλεκτρονικός έλεγχος. Έκλεισε η ψηφοφορία. 8 με 17 απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. 13 υπέρ. Ο κύριος Πιτέλα υπέρ. 14 υπέρ προς 10 εγκρίνεται. Οι 12 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Ja, 14. The vote is open. The vote is closed. Hm, everybody is against. Okay. 22 zu 1. Λοιπόν, 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. 23 με 24 είναι το αποτέλεσμα. Μισό λεπτό, διορθώνει η πρόεδρος. 25-0 εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Χίρς. Πολύ ωραία. jetzt kommen wir zu dem äh, Thema äh, Online Gambling. Λοιπόν, Skuria Online Gambling. Ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, ηλεκτρονικός τζόγος αν θέλετε. So, Bellet. Ja, bist kein Gambler. Bellet ist der Gambler. Okay. An die Arbeit. Λοιπόν, συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, γκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Η 3. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Η 36. Υπέρ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Η 5 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Μισό λεπτό, η 13 υπέρ. Α, θα το πω στα αγγλικά. Αγγλικά θα ψηφίσουμε. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Is closed. Ε, πέρας ψηφοφορίας. 15-9. Εγκρίνεται. Πιτέλα, κοιμάσαι. Είσαι κατά. Ε, πρέπει να μας δείξεις τι ψηφίζεις. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγγνώμη. Έκανα λάθος. 14 συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικός. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 26 0 συγχαρητήρια. Ποτέ δεν είδα τόσο σύντομη έκθεση με τόσο πολλές τροπολογίες. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε το αποτέλεσμα. Κύριε Πιτέλα, προσπάθησα να είμαι τόσο γρήγορη όσο εσείς χωρίς να μου λένε οι άλλοι μα πόσο γρήγορα πάτε, πόσο γρήγορα πάτε. Ποτέ δεν μπορεί να πάει κανεί αρκετά γρήγορα. Και ξέρω τώρα ότι θα διάσει η αίθουσα. Κύριε Αντιπρόεδρε, φεύγετε. Καλά. Πάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Bon, alors, wir können jetzt nicht zu Punkt 10 gehen, weil der Berichterstatter wahrscheinlich... Δεν μπορούμε να περάσουμε στο 10, διότι από ό,τι φαίνεται ο εισηγητή ε, δεν είναι ακόμα εδώ. Πάμε στο 11. Ούτε και αυτό είναι εδώ. Α, τι να πω κι εγώ. Η κυρία Τρούπελ είναι πάντα εδώ. Πάμε στο 12. <clears throat> Η κυρία Τρούπελ, παρακαλώ. Ε, η Χέλγα. Ευχαριστώ πολύ, Ντόρις. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Λοιπόν, εφόσον έχουμε μιλήσει γενικά για την προσέγγιση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το πώς ακριβώς ε, φαντάζεται το μέλλον ε, της, των εταιριών αξιολόγησης λογικών δικαιωμάτων, τώρα βρισκόμαστε στη φάση των τροπολογιών τις τελευταίες εβδομάδες. Είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις και εκτός από τις ε, τροπολογίες που ε, σας υπέβαλα έχω και μία αιτιολογία για το πώς ακριβώς σκέπτομαι όλα αυτά τα θέματα και τι θέλω να επιτύχω πολιτικά. Και έτσι λοιπόν ε, θέλω να σας παρουσιάσω κάποιες βασικές μου απόψεις. Για μένα λοιπόν υπάρχει η μεταρρύθμιση των ε, εταιριών αυτών στο πλαίσιο της ε, πολιτισμικής ε, πολυμορφίας. Αυτό είναι πάντα ο στόχος μας, κυρίως εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού, αλλά πρέπει να πω ότι όλα αυτά αναφέρονται και στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Άρα δηλαδή πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι προτάσεις. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στις τροπολογίες μου και επίση, και όσον αφορά την ε, προσπάθεια μεταρρύθμιση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλω να σα πω ότι τα τελευταία χρόνια οι εταιρείε αυτές ε, υπάρχουν ε, σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, οι οποίες εταιρείε όμως αυτές δεν έχουν δουλέψει τόσο ε, με τέτοια μεγάλη ακρίβεια όπως θα το επιθυμούσαμε. Παραδείγματο χάρη, στην ε, Ισπανία έχουν υπάρξει ε, δύσκολες περιπτώσεις, έχει προκύψει πολλές φορές και διαφθόρα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιους όρους που θα καθιστούν αδύνατο κάτι τέτοιο. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι θα πρέπει να δούμε λιγάκι και τον ψηφιακό κόσμο. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι να ασχοληθούμε με τις μεταρρυθμίσεις για να αλλάξουν και οι εταιρείε αυτές. Η ε, σημασία όλων αυτών δεν αμφισβητείται του αντίον περισσότερο από ότι το πράττει η Επιτροπή. Εγώ θα ήθελα να τονίσω τον ειδικό χαρακτήρα εταιριών ε, για την συλλογική διεκδίκηση δικαιωμάτων. Γιατί εδώ Πρόκειται για εταιρείε οι οποίες ε, λειτουργούν στην αγορά, όμως δεν είναι οργανώσεις, ε, γνήσιες οργανώσεις αγοράς. Δηλαδή έχουν τις ίδιες ε, ταρίφες για τους καλλιτέχνες, είτε είναι mainstream είτε όχι. Και αυτή λοιπόν η προσέγγιση η οποία διαφωνεί και αντιβαίνει σε μεταρρύθμιση όλων των ε, δικαιωμάτων. Αυτό θέλω να το διατηρήσω. Νομίζω όμως ότι σε πολιτικό επίπεδο υπάρχουν και ιδιωτικέ εταιρείε, δεν θέλω βέβαια να τις αναφέρω, οι οποίες εταιρείε αυτές έχουν τελείως ε, διαφορετικά συμφέροντα και θα επιθυμούσαν να εκμεταλλευτούν τα δικαιώματα των ε, επιτυχημένων καλλιτεχνών στην αγορά. Βεβαίως αυτό αντιβαίνει στις στη φύση των εταιριών αυτών που έχουν μια πιο δίκαιη προσέγγιση. Ο δικός μου λοιπόν ο στόχος ε, είναι αυτές τις ε, εταιρείε ε, να τις διατηρήσουμε, να καταστήσουμε σαφές γιατί έχουν μια ιδιαιτερότητα και γιατί σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχουν κονδύλια που διοχετεύονται στην προαγωγή, των, στην στήριξη των νέων στην εκπαίδευση και αυτή η βασική λειτουργία των εταιριών ε, συλλογικής άσκησης ε, δικαιωμάτων ε, αυτές πράγματι αγωνίζονται για, την, για τον πολιτισμό, για την πολυμορφία, για τους καλλιτέχνες οι οποίοι ε, πολύ συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες γιατί δεν είναι όλοι τόσο επιτυχημένοι όσο η Μαντόνα. Εγώ λοιπόν ε, θέλω να διαφυλαχθούν όλα αυτά και ακριβώς αυτός είναι ο στόχος μιας τροπολογίας μου. Δηλαδή τα κράτη-μέλη να μεριμνήσουν έτσι ώστε οι εταιρείε ε, συλλογικών δικαιωμάτων να προβλέψουν τέτοιου είδους κονδύλια. Και αυτό δεν προβλέπεται με απόλυτη σαφήνεια στην πρόταση της Επιτροπής και θα ήθελα να το αλλάξω. Γνωρίζετε λοιπόν ότι συλλογικά υπάρχει μια αντιπαράθεση σχετικά με την, με την οδηγία παροχής υπηρεσιών ε, που βέβαια είναι και νόμος και δεν αμφισβητείται, παρόλα αυτά σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει μία αντιπαράθεση για το κατά πόσον οι εταιρείε αυτές ε, συλλογικών ε, δικαιωμάτων, κατά πόσον οι εταιρείε αυτές ε, μπορούν να την χάνουν πλήρους υποστήριξης. Αυτές λοιπόν οι εταιρείε εξαιρέθηκαν από την οδηγία περί παροχής υπηρεσιών. Υπάρχει λοιπόν μια αντιπαράθεση που σοβεί εδώ και πολλά χρόνια και δεν νομίζω ότι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ισχύει απλά και μόνο η οδηγία περί παροχής υπηρεσιών. Πρέπει να δούμε λιγάκι ποια είναι αυτή η ιδιαιτερότητα αυτών των ε, εταιριών. Και κατόπιν τούτου όλα αυτά εγώ τα αναφέρω στο αιτιολογικό της εκθεσής μου για να καταστήσω απόλυτα σαφές ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ε, καθαρόεμες ε, εταιρείε της αγοράς. Το επόμενο σημαντικό θέμα είναι το εξής. Στις επιγραμμικές αδειοδοτήσεις και γι' αυτό τον λόγο κάνει και η Κομισιόν αυτή την πρόταση. Ε, στην αρχή μιλάει για διαφάνεια. Το δεύτερο τμήμα της οδηγίας αναφέρεται στην επιγραμμική αδειοδότηση, αλλά μόνο σε ε, μουσικά κομμάτια. Θα ήθελα λοιπόν, εκτός από αυτές τις ε, εταιρείες ε, συλλογικών δικαιωμάτων, θα ήθελα να υπάρχουν και ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες και αυτές όμως θα υπόκεινται στις διατάξεις περί διαφάνειας. Γιατί αλλιώς ε, φοβάμαι ότι αυτές οι εταιρείες ε, θα δεσμεύονται με κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Αν όμως άλλες εταιρείες δεν υπόκεινται στους ίδιους αγώνες, αυτομάτως ε, προκύπτει ε, στρέβλωση του ανταγωνισμού. Γιατί οι εταιρείες ε, οι συλλογικών δικαιωμάτων θα έχουν τελείως, διαφορετικές, τελείως διαφορετικούς όρους με τους οποίους θα λειτουργούν. Εγώ όμως δεν είμαι κατά του ανταγωνισμού, είμαι υπέρ του θεμητού ανταγωνισμού. Αυτοί λοιπόν οι κανόνες είναι σημαντικοί για να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός και εδώ στηρίζω την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι δημιουργοί πρέπει να έχουν οι τη δυνατότητα να επιλέγουν μόνοι τους τις εταιρείες ε, που θα τους ε, εκπροσωπούν, ίσως να θέλουν να συνεργαστούν με εταιρείε εκπροσώπησης ε, και σε άλλες χώρες, εφόσον αυτό το κρίνουν προσιτό και ενδιαφέρον. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα και είμαι σίγουρη ότι επ' αυτού θα έχουμε κάποια αντιπαράθεση. Εγώ προσωπικά επιθυμώ οι δημιουργοί να έχουν τη δυνατότητα με μονομένα έργα να τα αποσπούν από τις εταιρείε και ε, να τα προβάλλουν μόνοι τους. Γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια μιλάμε για τα δικαιώματα του δημιουργού και προσπαθούμε να βρούμε κάποια ισορροπία. Ξέρετε ότι αυτή είναι η δική μου η προσέγγιση. Αφενός ε, θεωρώ ότι πρέπει οι δημιουργοί να αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα στο σημερινό ψηφιακό κόσμο. Παράλληλα όμως ε, θα πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα επιλογής. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, να μπορούν να δουλεύουν με ελεύθερες άδειες. Αυτό δεν αντιβαίνει στους κανόνες περί δικαιωμάτων δημιουργού, αλλά παρόλα αυτά ανοίγει νέες ευκαιρίες. Αυτή λοιπόν είναι μια προσέγγιση την οποία έχω συμπεριλάβει στις τροπολογίες που έχω καταθέσει. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για μένα. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τις ε, άλλες ε, τροπολογίες, ε, προσπαθώ όπου κατά την άποψή μου κρίνω ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια, να το προβάλλω αυτό. προσπαθώ να πω ότι τόσο οι χρήστες όσο και οι πελάτες να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ψηφιακές δυνατότητες, την πρόσβαση σε δεδομένα. Βεβαίως ε, δεν θα πρέπει να είναι προσωπικά τα δεδομένα που θα εμπίπτουν στην προστασία ιδιωτικών δεδομένων. Παράδειγμα, ας πούμε, ε, εάν υπάρχουν έργα τα οποία εμπίπτουν στον δημόσιο τομέα, Αυτά τα έργα έχουν ε, πληροφορίες που μπορούν να ε, διατεθούν, όχι όμως ε, ατομικά δεδομένα για τον δημιουργό. Αυτά αφορούν καθαρά και μόνο τον δημιουργό και αυτά πρέπει να προστατεύονται από τις εταιρείε. Αυτά ε, έτσι σε γενικές γραμμές όσον αφορά στην προσέγγιση μου και κατά τα άλλα χαίρομαι πάρα πολύ που τις αμέσως επόμενες εβδομάδες θα έχουμε συνεργασία. Χαίρομαι και για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει και που θα ακούσω την κριτική σας και τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Χέλγα, λέει πρόεδρος. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί συνεχώς ε, τα τελευταία χρόνια γιατί έχουμε πάρα πολλούς ε, που έρχονται σε εμά και περιμένουν τη βοήθειά μας. Ε, νομίζω λοιπόν ότι στον τομέα αυτό μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί ένα πράγμα είναι απόλυτα σαφές. Δεν μπορούν όλα αυτά να βρίσκονται στα χέρια αυτών των εταιριών και όταν ε, ε, βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών να μην υπάρχει διαφάνεια. Ο κύριος Καβαντά έχει ζητήσει το λόγο. Ντόρις, αγαπητοί συνάδελφοι, Κυρίε και κύριοι, μπορούμε να ευχαριστήσουμε την Έλγα για μια πάρα πολύ εξαιρετικά ισοσχελισμένη έκθεση με την οποία συμφωνώ σε γενικές γραμμές. Βεβαίως θεωρώ ότι αυτές οι εταιρείε συλλογικών δικαιωμάτων είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν την σωστή κατανομή των δικαιωμάτων σε αυτούς που τα δικαιούνται. Να υπενθυμίσουμε πώς έχουν το θέμα αυτό. Από την ε, ερμηνεία των έργων των δημιουργών απορρέουν δικαιώματα τα οποία ε, συλλέγουν και κατανέμουν αυτού του είδους οι εταιρείε. Έτσι πρέπει να λειτουργεί το σύστημα. Και δικαίως επιμένεις ότι θα πρέπει ε, να υπάρχει διαφάνεια. Και στη χώρα μου. Η σωστή κυβέρνηση και διαφάνεια κάποια χρόνια πριν δεν ήταν ε, σωστή. Και πρέπει να το πούμε αυτό με απόλυτη ευκρίνεια. Αυτές οι εταιρείες, οι ιδιώτες, οι εμπορικές επιχειρήσεις όπως είπες, θα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες διαφάνεια με αυτό που έχουν και όλες οι εταιρείες ε, ε, συλλογής τέτοιου είδους δικαιωμάτων. Δεδομένου ότι εδώ έχουμε χρήμα που δεν τους ανήκει, αλλά ανήκει στους δημιουργούς. Είμαι, όπως και εσύ, πεπισμένος ότι ο κατακαιρματισμός αυτών των δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει σε όλες τις διαδικασίες πολύπλοκες και δημιουργεί άχθος ε, και αυξάνει το κόστος για αυτούς που δικαιούνται χρήματα. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν αυτών των εταιριών που κυρίως ε, έχουν σχέση με τα οπτικοακουστικά συστήματα και τις, ε, τις ε, απευθείας μεταδόσεις και τις τα ζωντανές μουσικές παραγωγές είναι κάτι το διαφορετικό, θα πρέπει να έχει κανόνες και βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι υπάρχουν και μη ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει εκεί επίσης να εφαρμόζονται τα ίδια δικαιώματα για να μην καταστρατηγούν τα δικαιώματα των δημιουργών και να λάβουν υπόψη για το τι γίνεται στο ίντερνετ. Λυπούμε διότι στην πρόταση οδηγίας εξομοιώνονται αυτές οι εταιρείες με παρόχους υπηρεσιών σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει το άρθρο 4.1 της οδηγίας για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ο στόχος αυτών των εταιριών δεν είναι να αναπτύξουν μια εμπορική δραστηριότητα, αλλά να κάνουν ε, την διαχείριση δικαιωμάτων, να τα καταμείνουν, να κατανείμουν και να κάνουν ε, δραστηριότητες ε, ε, κοινού δημοσίου ενδιαφέροντος. Άρα δεν δημιουργούν κέρδος και δεν θα πρέπει να ε, καταλήγουν σε επενδύσεις οι οποίες μπορούν να αποβούν καταχρηστικές. Τώρα, δεδομένου ότι εδώ δεν έχουμε ως στόχο το κέρδος, θα πρέπει να μπορούν οι εταιρείε αυτές να επενδύουν το ενεργητικό τους με τρόπο που δεν θα δημιουργεί κίνδυνο σε όλα αυτά τα προϊόντα που θέλουν να διασφαλίσουν, δηλαδή τα δικαιώματα των ε, μουσικών, δημιουργών, συγγραφέων κτλ. Επίσης ε, αναφέρεται εδώ την χρονική περίοδο των ε, τριών ετών. Ίσως μπορούμε να διαφοροποιηθούμε όσον αφορά το χρόνο με τον οποίο θα πρέπει να δοθούν τα δικαιώματα. Αν ξεπεραστεί αυτός ο χρόνος, ίσως θα πρέπει τα κέρδη που υπάρχουν, τα δικαιώματα δηλαδή, σε χρήμα, να επενδυθούν στον ε, τομέα των πολιτιστικών για κοινωνικό θέματα. Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε κατάχρηση, διότι μπορεί να υπάρξει στον τομέα αυτό πολύ συχνά, θα πρέπει από νομικής πλευράς να ε, μειώσουμε τις, ε, τα δικαιώματα και τις εξουσίες που έχουν ε, γενικές ε, συνελεύσεις οι οποίες μπορεί να αποτελούνται από ελάχιστα άτομα που έχουν στο χέρι τους όλη τη δύναμη και μπορεί να καταλήξουν σε δυσάρες καταστάσεις. Ε, το έχουμε δει αυτό. Επίσης πρέπει να πω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να βοηθήσουμε τους δημιουργούς, να προστατεύουμε τα δικαιώματά τους, να λαμβάνουμε υπόψη επίσης τις μικρές και μεσές τέτοιου είδους εταιρείες και κυρίως να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των δημιουργών. Διαρωτώ με, μήπως δεν θα πρέπει να υπάρξει μία αρχή διαβούλευσης και επιτήρησης της διαφάνειας για αυτές τις ε, εταιρείε είναι ιδιωτικέ 100% ή είναι ένα συνδυασμός ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή να κάνουμε ένα κάποιο ίδρυμα ο οποίος ε, να μπορεί να ελέγχει την όλη κατάσταση ώστε να μην έχουμε καταχρήσεις εις βάρος των δημιουργών. Αυτά ήθελα να πω και πάλι συγχαρητήρια και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Ζων Μαρή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και την Χέλγα. Ε, Νομίζω γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό ήταν ένα Ηράκλειο έργο. Και πολύ καλές λοιπόν οι προτάσεις που κατέθεσες ε, και ε, νομίζω ότι πρέπει να ε, βρούμε σύντομα κάποια συμφωνία και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να χαιρετήσουμε την προσέγγιση της ε, Κομισιόν, δηλαδή όσον αφορά αυτές τις εταιρείε εκπροσώπησης να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Όλοι μας βέβαια διαπιστώσαμε ότι όταν τα είδαμε αυτά πιο προσεκτικά ότι υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια με την έννοια ότι οι κανόνες ε, για τις ε, εταιρείες αυτές υπάρχουν. Από την άλλη όμως υπάρχουν και άλλες ε, εταιρείες στην αγορά Κατόπιν τούτου για αυτές τις ε, εταιρείε ε, εκπροσώπησης πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, η οποία διαφάνεια όμως ε, δεν ισχύει με τον ίδιο τρόπο για μουσικές εταιρείε. και νομίζω αυτό είναι ένα πρόβλημα, το είπες και εσύ. Αυτό είναι πρόβλημα ότι πλέον δεν υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός, άρα δηλαδή πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε σε ένα σύστημα όπου οι εταιρείε αυτές ε, κατά κάποιον τρόπο ε, είναι και συνδικαλισμένες μεταξύ τους και ε, διαφυλάσσουν τα δικαιώματα των εταιρείων, αυτές ενδέχεται κατά κάποιον τρόπο να παρακαμφθούν. Δηλαδή όλοι οι δημιουργοί να απευθύνονται στις ιδιωτικές εταιρείε και οι εταιρείε εκπροσώπησης να παίρνουν μόνο τα υπόλοιπα, τα ψίχουλα. Και αυτό είναι πρόβλημα όχι μόνο για τους καλλιτέχνες, αλλά και για τον, ε, ε, την πολιτιστική εκπροσώπηση. Δηλαδή οι εταιρείε αυτές ε, να μην είναι οργανωμένες με κριτήρια αγοράς, αλλά ε, να έχουν κάποια άλλη μορφή οργάνωσης και να αδικούνται. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο σημείο αυτό να προσέξουμε όσον αφορά στις ε, τροπολογίες. Το άλλο πρόβλημα το σε ε, πρόκειται για την οδηγία παροχή υπηρεσιών, κατά πόσο ισχύει ή όχι. Και αυτό πραγματικά είναι παράδοξο. Από τη μια οδηγία παροχής υπηρεσιών ε, λέει ότι τα δικαιώματα του δημιουργού δεν συμπεριλαμβάνονται ε, σε αυτήν την οδηγία. Από την άλλη όμως ε, συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείε που εκπροσωπούν τους δημιουργούς. Πολύ περίεργα τα πράγματα. Και κατόπιν τούτου θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι εδώ δεν μιλάμε για εμπορεύματα αλλά για ένα πολιτιστικό αγαθό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ιδιωτικές εταιρείες ε, και αυτές ε, πρέπει να υπόκεινται σε κάποιους ε, κανόνες διαφάνειας. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ε, ε, και θα πρέπει οι εταιρείε να οργανώνουν συναντήσεις διοικητικού συμβουλίου. Ε, και θα πρέπει να ισχύουν κανόνε ε, διαφάνειας για να αποφεύγεται ο ανταγωνισμός. Ε, κατά την άποψή μου αυτό είναι απολύτω απαραίτητο, πολύ σημαντικό. Κατόπιν τούτου ίσω μπορούμε, όπως είπε και εσύ, σε κάποια σημεία να κάνουμε καλύτερο έλεγχο να είμαστε λίγο πιο σαφείς. Ε, καταρχήν όμως ε, συμφωνούμε και νομίζω ότι τελικά ε, θα έχουμε πολύ καλή βάση για την συνέχιση των εργασιών μας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η κοινωνική ευθύνη την οποία αναλαμβάνουν οι εταιρείε εκπροσώπησης που αναλαμβάνουν να προάγουν τα πολιτιστικά αγαθά. Αυτό να αναφέρεται με απόλυτη σαφήνεια ε, κυρίως ε, για τις εταιρείε που δεν το κάνουν. Αυτά όλα τα βρίσκω πάρα πολύ λογικά, σημαντικά, γιατί με τον τρόπο αυτό ε, οι εταιρείε αυτές κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Και το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Πέτρα, η Σαμπίνε. Καταρχήν θα ήθελα να στηρίξω πάρα πολλά από αυτά που είπε η Helga Τρούπελ. Νομίζω ότι αναφέρθηκαν πολλά και σημαντικά σχετικά με την σημασία των εταιριών εκπροσώπησης ε, για τον ε, πολιτιστικό τομέα. Εγώ στηρίζω αυτή την τάση για περισσότερη διαφάνεια. Νομίζω ότι ανάμεσα στις διάφορες εταιρείε εκπροσώπησης υπάρχουν πολλές διαφορές. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αναφέρονται κάποιες ε, ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά τη διαφάνεια. Για μένα μικρό πρόβλημα είναι αυτή η σχέση ανάμεσα σε ιδιωτικές εταιρείε, πρακτορία, δηλαδή και εκεί να υπάρχει η ίδια διαφάνεια όπως και για τις εταιρείε, αυτό που απαιτούμε. Ε, δύσκολο αυτό, σε τελική ανάλυση όμως ε, εδώ πρόκειται για μια καθαρή σύμβαση ανάμεσα σε εντολοδόχο και εντολέα. Άρα δηλαδή θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο την, ε, την κατάσταση αν ισχύουν ίδιες προδιαγραφές. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν μεγαλύτερη διαφάνεια. Εγώ επίσης ε, στηρίζω πλήρως αυτά που ελέγχθηκαν σχετικά με την ε, οδηγία παροχής υπηρεσιών. Θεωρώ ότι εδώ έχουμε ένα καθήκον το οποίο είναι πολύ ευρύτερο από το να προσφέρεται απλά ε, μία υπηρεσία. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα αυτό το οποίο κατέθεσε η Κομισιόν νομίζω ότι κατά την άποψή μου ε, δεν στέκει. Τώρα, κάτι που κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό είναι το θέμα των ε, αδειοδοτήσεων, το δεύτερο που θίγεται στην ε, οδηγία. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια για να μπορούμε να ε, θέτουμε σε ισχύ αυτές τις αδειοδοτήσεις πολλαπλής εδαφικής ισχύω. να είναι βέβαια διαφανής η συνεργασία. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Και αυτό αποτελεί μια σημαντική βάση όχι μόνο ε, για τους ε, δημιουργούς ε, αλλά και για τους χρήστες. Να υπάρχει μια τράπεζα δεδομένων όπου να αναφέρεται πώς ακριβώς εκπροσωπούνται αυτοί, έτσι ώστε ως χρήστης άδεια να έχει κανείς πρόσβαση και να μπορεί και ο ίδιος να φέρεται νομότυπα. Γνωρίζω ότι επ' αυτού εργάζονται αρκετές εταιρείε εκπροσώπησης. Βεβαίως πρέπει να πω ότι ε, δεν έχουμε επιτύχει απόλυτα το στόχο μας. Άρα δηλαδή αυτό να το προβάλλουμε ότι χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Διότι θεωρώ ότι το θέμα των εταιριών εκπροσώπησης πρέπει κανείς να το δει από δύο σκοπιές. Αφενός ε, από την πλευρά ε, των ε, δημιουργών που ε, θέλουν να εκπροσωπούν σωστά τα δικαιώματά τους. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό το ότι οι εταιρείε εκπροσώπησης δεν είναι απλά εταιρείε για να συγκεντρώνουν κεφάλαια, υπάρχουν για να εκπροσωπούν τα δικαιώματα. Θεωρώ λοιπόν αυτό ισχύει και από την άλλη πλευρά είναι σημαντικό κάποιος που επιθυμεί να αποκτήσει μια άδεια για να χρησιμοποιήσει ένα έργο ε, να μπορεί να το επιτύχει αυτό με ταχύτητα και διαφάνεια ε, και όχι να παίρνει διπλούς και τριπλούς ε, λογαριασμούς από διάφορες εταιρείες διότι ενδεχομένως να υπάρχουν δικαιώματα που εκπροσωπούνται δύο και τρεις φορές. Όλα αυτά να είναι σαφέστερα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 Market Committee, and the two will very much feed into what's happening in jury. Thank you. Vielen Dank. Ich hätte gerne noch gewusst, äh, Helga. Πρόεδρος, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Helga. Εφόσον προτείνουμε να συσταθούν παντού αυτοί οι οργανισμοί και αυτά τα ταμεία, ε, τελικά τι θα γίνει με τα χρήματα ε, πώς ακριβώς θα επιμερίζονται τα κονδύλια και ποιος ε, θα είναι ο αποδέκτης αυτών των κονδυλίων. Ε, γιατί υποτίθεται ότι θα αποφελούνται όλοι ή μήπως θα αποφελούνται μόνο όσοι έχουν ενταχθεί σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν δεν ζητάει κανείς το λόγο θα δώσω το λόγο στην Χέλγκα και μετά στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους. Σε γενικές γραμμές νομίζω συμφωνείτε με την έκθεσή μου. Βέβαια ασκήσατε και κάποια κριτή. Θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπε ο κ. Καβαντά. Ότι ε, καταρχήν επιθυμεί τον ε, θεμητό ανταγωνισμό. Βεβαίως και εγκρίνει αυτούς τους ε, οργανισμούς ε, συλλογικής διαχείρισης ε, και εγώ συμφωνώ με αυτό. Η Πέτρα τόνισε ότι ε, τα δικαιώματα των γραφείων θα πρέπει και αυτά να υπόκεινται στην διαφάνεια. Αναφέρθηκε επίση ότι πρέπει να δούμε λιγάκι αυτές τις ιδιωτικέ συμβάσεις ε, ε, και κατά πόσον ισχύουν ε, οι κανόνες διαφάνειας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πολιτικά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επικρατεί διαφάνεια. Διότι αλλιώ, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, είναι σαφές ότι θα υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αυτό θα πλήξει κυρίως ε, τους λιγότερο επιτυχημένους καλλιτέχνες. Εμείς όμως επιθυμούμε η πολιτιστική πολυμορφία να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, να διαφυλάσσετε ως αγαθό. Κατόπιν αναφέρθηκαν και κάποια άλλα στοιχεία για το μεγάλο ενδιαφέρον ε, που έχουμε ε, σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού. Νομίζω πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Τα κέρδη, τα ε, χρήματα που δικαιούνται να τους διατίθενται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αυτό λέχθηκε και συμφωνώ με όλα αυτά. Κατόπιν, μια άλλη ιδέα που αναφέρθηκε είναι η εξή. Κυρίως σήμερα που υπάρχουν ψηφιακές δυνατότητες, ε, το να υπάρχουν τράπεζες δεδομένων όπου όλοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ε, τράπεζες και οι χρήστες ε, και οι δημιουργοί. Επειδή υπάρχουν όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη αποζημίωση των δημιουργών, αλλά θα πρέπει να προσφέρονται και περισσότερες πληροφορίες και στους χρήστες ε, και στους ε, δημιουργούς, κυρίως σχετικά με την αδειοδότηση. Όσον αφορά στους ε, οργανισμούς ε, συλλογικής διαχείρισης, ε, θα πρέπει να τονίσουμε ότι όταν υπάρχουν δίκαιοι κανόνες σχετικά με την αδειοδότηση, νομίζω ότι μπορούν καλύτερα να προστατευτούν τα έργα του δημιουργού. Η Έμα Μακλάκιν με χαροποίησε αυτό υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι η περαιτέρω εξέλιξη της ψηφιακής κοινή αγοράς και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Οτιδήποτε κάνουμε τελικά πρέπει να αποβλέπει στον υπάρχει λειτουργικότητα και όχι εμπόδια. Και είπατε επίσης ε, ότι όσον αφορά αυτούς τους οργανισμούς ε, συλλογικής διαχείρισης ε, θα πρέπει να οριστούν καλύτερα αυτοί οι οργανισμοί. Χαίρομαι πάρα πολύ που στηρίζετε την πρότασή μου. Και βέβαια είπατε όλοι ότι θα καταθέσετε προτάσεις βελτίωσης. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Για οτιδήποτε ε, γίνει σαφέστερο και αποτελέσει βελτίωση, νομίζω ότι αυτό συμφέρει όλους μας. Και όσον αφορά την τελευταία ερώτηση της κυρίας Πακ, πράγματι αυτά τα ταμεία που υπάρχουν για τον πολιτισμό και την κοινωνική εξασφάλιση των καλλιτεχνών αφορούν κυρίως ε, τους, ε, τα μέλη των οργανισμών συλλογική διαχείρισης και τους νέους καλλιτέχνες. Είναι λοιπόν εργαλεία ε, που αποβλέπουν στο ευρύτερο κοινό καλό στον τομέα του πολιτισμού γιατί θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστούν καλύτερα οι καλλιτέχνες, κυρίως οι νέοι. Αυτό κάποιες ιδιωτικές εταιρείε δεν το κάνουν. Αυτές ε, αποσκοπούν στο κέρδος, εκμεταλλεύονται τους καλλιτέχνες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεν επενδύουν όμως σε νέους καλλιτέχνες και σε πολιτιστική πολυμορφία. Το να υπάρχει όμως αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό γιατί όλοι μας τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε κάνει την εμπειρία μας με ε, εταιρείε που είναι πάρα πολύ καλές ε, στην ε, εκπροσώπηση, όχι όμως στις επενδύσεις. Για μένα οι εταιρείε της οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης διαδραματίζουν ένα πολύ συγκεκριμένο κοινωνικό ρόλο που όμως δεν λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία σε μεγάλο βαθμό ε, κατά αυτών των οργανισμών. Ξεχνάει όμως ότι αυτοί οι οργανισμοί έχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο. Δεν μπορούμε σε όλες τις περιπτώσεις να λέμε αν ναι, εδώ αυτό είναι μονοπόλιο και εκεί τελειώνει. Θα πρέπει να δει κανείς λιγάκι τους οργανισμούς συλλογική διαχείρισης, πώς μπορούν να βελτιωθούν χωρίς να καταστρέψει κανείς αυτά που προσφέρουν στο ευρύτερο κοινό. Αυτή είναι η πολιτική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Η κυρία Φονχάιν ε, κατέστησε σαφές ε, τι ακριβώς συμβαίνει με την εφαρμογή της ε, οδηγίας παροχής υπηρεσιών και γιατί σε αυτή την περίπτωση, επειδή πρόκειται για ιδιαίτερα δικαιώματα, γιατί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες ε, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία, βεβαίως και αργότερα και σε συνεργασία με άλλους ε, συναδέλφους. Εάν λοιπόν ε, κατορθώσουμε αυτόν τον ρόλο της πολιτιστικής πολυμορφίας να τον προβάλλουμε, θα επιτύχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και ε, ίσως περάσουμε και την έκθεσή μας στην Ολομέλεια. Θα χαρώ πάρα πολύ. Και εμείς θα χαρούμε, λέει η Πρόεδρος, και γι' αυτό σας παρακαλώ τις τροπολογίες να τις καταθέσετε μέχρι τις 14 ε, Μαΐου. Υπάρχει αρκετός χρόνος για να τα σκεφτείτε όλα αυτά. 14 λοιπόν Μαΐου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα μέχρι το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε την Χέλγα. Μισό λεπτό, ε, ξέχασα την... Ε, Επιτροπή, την κυρία Μαρτίν Πχάτ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, Madam Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και συγγνώμη, διότι έφτασα στο μέσο της συζήτησης. Νόμιζα ότι προβλεπόταν η συζήτηση 10.30. Εν πάση περιπτώσει, μπορώ να τρέξω αρκετά γρήγορα, αλλά όχι πιο γρήγορα από ό,τι μπορώ από το γραφείο μου. Αρχίζοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Τρούπελ, για την έκθεσή της και κυρίως για τις προσπάθειες που κατέβαλε ώστε να κάνει διάλογο, να υποβάλει ερωτήσεις και να κατανοήσει το όλο θέμα. Έχουμε λοιπόν να εκφράσουμε το βασμό μας για το πόσο εμπεριστατωμένη είναι η έκθεσή της. Συμφωνούμε με κάποιες τροπολογίες, με όχι, αλλά εν πάση Τώρα, για κάποια θέματα τα οποία τέθηκαν εδώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα πω το εξή. Πολύ σύντομα, ας, ας εξηγήσω ποια είναι η λογική η οποία άπτεται τις οδηγίες αυτή. Είναι πολύ βασική. Η επιλογή των κατόχων δικαιωμάτων. Πιστεύουμε ότι οι δημιουργίες τις οποίες χειρίζονται τέτοιου οργανισμοί διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων πρέπει να είναι της επιλογής των δημιουργών. Αυτοί λοιπόν οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πρέπει να έχουν την ε, ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για το πώς θα χειριστεί κανείς τα δικαιώματά τους. Και η καλλιτεχνική και η πολιτιστική πολυμορφία υπάρχει μόνο όταν μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή η πολυμορφία. Δεν ακούτε? Δεν ακούτε? Δεν με ακούτε τώρα? Για Μας ακούτε? Συγγνώμη. Για τις δημόσιες αρχές. Υπάρχουν ε, διάφορα στοιχεία τα οποία έχετε θέσει υπήρχαν αναφορές σε σχέση με το κατά πόσο θα έπρεπε να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για όλους. Σωστό είναι αυτό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και ποιοι άλλοι δεν, κάποιοι δεν έχουν το, το ίδιο είδος δραστηριότητες. Ε, μερικές φορές κάποιοι είναι agents, ε, είναι διαφορετικό πράγμα ε, να μιλάμε για οργανισμό συλλογική διαχείρισης και για τους agents. Είναι πολύ σημαντικό αυτό υπάρχουν και ενδιάμεση στην αγορά αυτή. Υπάρχουν ορισμένες φορές ε, και μονοπόλια. Συνήθως ε, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ζητούν ε, αποκλειστική εντολή από τα μέλη τους. Κάποιοι άλλοι οργανισμοί δεν το κάνουν. Είναι πράγματα λοιπόν που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Υπήρξε μία συζήτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει βεβαίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελε να το κατανοήσει καλύτερα. Κάτι ακόμη η καλύτερη διανομή. Πράγματι, απολύτως συμφωνούμε, θα έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και καλύτερη η διανομή και συντομότερη, όμως πρέπει να είναι και ακριβής. Είναι πάρα πολύ εύκολο να διανύμει κανείς ε, γρήγορα από το να διανύμει σωστά. Λοιπόν, ορισμένα, ορισμένες από τις διαδικασίες μπορεί να φαίνονται χρονοβόρες, αλλά μερικές ε, φορές ε, είναι απαραίτητος αυτός ο χρόνος ε, για να φτάσουν τα χρήματα στο σωστό καλλιτέχνη, στον κάτοχο των δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που προσπάθησε να κάνει είναι να προωθήσει την ιδέα αποτελεσματική ε, ε, ε, πλήρους ε, ενημερωμένης βάσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Το κατά πόσο τώρα αυτό θα είναι ε, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τίποτα στους οργανισμούς αυτούς. Μπορούμε να τους υποχρεώσουμε να έχουν τα σωστά εργαλεία, αλλά τώρα τι μορφή θα πάρουν αυτά τα εργαλεία. Υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσει στην αγορά, το γνωρίζετε αυτό. Είναι δύσκολο να το επιβάλλουμε αυτό μέσω νομοθεσία στους οργανισμούς. Κάτι ακόμη και θα ολοκληρώσω είναι το ισότιμο πεδίο για όλα τα κράτη-μέλη. Κοιτάξτε, Σωστό είναι αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν το συζητούμε αυτό. Κάποια είδη ελέγχου των οργανισμών ε, είναι καλύτερα από άλλα. Υπάρχει μια συζήτηση κατά πόσο ο καλύτερος τρόπος ελέγχου είναι να υπάρχει πρώτερη αδειοδότηση ή όχι. Η οδηγία έχει αποφύγει την επιβολή στα κράτη-μέλη την πρώτερη αδειοδότηση οργανισμών, δεν παρεμβαίνει με τα κράτη-μέλη που έχουν τέτοιο σύστημα και θέλουν να το διατηρήσουν. Γιατί ο βασικός λόγος είναι γιατί δεν είναι σαφές. Δεν είναι σαφές ότι το σύστημα της πρώτερης αδειοδότησης είναι αυτό, το, αυτό που θα λειτουργήσει καλύτερα σε όλα τα κράτη-μέλη. Αν δει κανείς ε, τον αριθμό των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης... Ε, ε, για παράδειγμα στι σκανδιναβικέ χώρε, δεν υπάρχει υποχρεωτικά το σύστημα τη πρώτερη αδειοδότηση, εκτό αν υπάρχει ειδική μορφή αδειοδότηση. Ε, Υπάρχουν περιπτώσεις πολύ καλής διαφάνειας, δεν θα πω συγκεκριμένα ονόματα γιατί δεν είναι κάτι το οποίο θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει, δεν μας αρέσει να το κάνουμε αυτό. Υπήρχαν περιπτώσεις μεγάλων προβλημάτων ε, με τη συμπεριφορά των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και τη διαχείριση των, των ε, ε, κεφαλαίων και υπήρχαν περιπτώσεις πρώτερης αντιδότησης από τις δημόσιες αρχές, ε, πρώτερης, πρώτερου ελέγχου από, τα, από τις αρμόδιες αρχές. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σημαντικό ρόλο για αυτούς τους οργανισμούς, χρειαζόμαστε διαφάνεια και πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ε, στο οποίο τρόπος ε, ελέγχου, στο οποίο υπάρχει ένας ρόλος για το δικαστήριο, ένα ρόλο για τις αρχές ε, ανταγωνισμού, η εσωτερική αγορά διαδραματίζουν το ρόλο τους. Είναι σημαντικό να μην υπάρχει ένας χρυσός κανόνας, ο οποίος θα έπρεπε να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη και βέβαια τα πολιτιστικά ταμεία. Όπως γνωρίζετε, η πρόταση είναι ουδέτερη. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε με τα πολιτιστικά ταμεία που επιβάλλει η νομοθεσία. Υπάρχουν κάποιες μορφές συλλογής επιτρέπεται στον οργανισμό να αποφασίζει κατά πόσο κάποια από τα έσοδα μπορεί να πηγαίνουν σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Δεν είναι υποχρεωτικό, είναι κάτι όμως το οποίο κατά τη γνώμη μας πρέπει να λαμβάνει ο ίδιος ο οργανισμός με τη συμμετοχή των μελών του. Αυτά ήθελα να πω σε γενικές γραμμές για τα σχόλια που άκουσα. Η Επιτροπή ως τώρα ε, όπως και πάντοτε παραμένει στη διάθεσή σας ε, και της εισηγήτριας και των ε, μελών της Επιτροπής σας για να συζητήσουμε αυτό το πολύ δύσκολο αλλά συναρπαστικό θέμα, η συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θέλω να σας πω το εξής, ότι προηγουμένως συζητήσαμε και βεβαίως δεν φταίτε εσείς ε, που δεν ήσασταν εδώ. Προχωρήσαμε γιατί αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη ως ε, αδαείς. Ε, λέω απλά ότι αυτά τα οποία συζητάμε δεν συμβαδίζουν με αυτά τα οποία έχουμε πει κατά το παρελθόν, αλλά σας είπα είμαι αδαίς λιγάκι σε όλα αυτά και θα δούμε στη συζήτηση και στις τροπολογίες ε, κατά πόσον θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση ή όχι. Ελπίζω λοιπόν ότι θα υπάρξει αγαστή συνεργασία ε, προ όφελο εκείνων των οποίων τα δικαιώματα επιθυμούμε να προστατεύσουμε. Ευχαριστούμε τη Χέλγα και πάμε τώρα πάλι πίσω στις ε, γλώσσες που απειλούνται. Κύριος Αλφόνση. Δεν είσαστε εσείς εισηγητής. Συνάδελφε Αλφονσί, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή μιλάει για την γλωσσική και πολιτιστική πολυμορφία που είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έκφραση της, ε, του πλούτου, του πολιτιστικού και γλωσσικού της Ευρώπης και συνεισφέρει και στον πλούτο της Ευρώπης. Ποιο είναι το πρόβλημα. Μπορούμε σήμερα να θεωρήσουμε ότι πολλές κουλτούρες και γλώσσες της Ευρώπης απειλούνται από εξαφάνιση. Από το 1996 στην UNESCO έγινε εξαιρετική δουλειά για να μπορέσουν να ευρεθούν τα επιστημονικά κριτήρια τα οποία θα μας ορίσουν πώς κάποιες ε, γλώσσες απειλούνται και πώς μπορούμε να βασιστούμε στο θεμελιώδες κριτήριο που είναι η μετάδοση από τη μια γενιά στην άλλη και πώς μπορούν οι γλω... κάποιες γλώσσες να αποδυναμωθούν διότι υπάρχει μία ισχύουσα. Τα κριτήρια αυτά ορίζονται με μεγάλη σαφήνεια και εξετώντας τα, τα, συγγνώμη, μπορούμε να δούμε ότι πάρα πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες σήμερα απειλούνται από εξαφάνιση. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, παντού, στην ε, Μεσόγειο, στον Ατλαντικό, στο Βορρά, κοντά στα Πυρηναία, καθώς και στην Κεντρική Ευρώπη και εκτός Ευρώπης βεβαίως, σε όλη την Ευρώπη και εκτός υπάρχει αυτή η κατάσταση που δημιουργεί πρόβλημα θεμελιώδους σημασίας για την διασφάλιση της πολυμορφίας και για την διασφάλιση αυτής της κληρονομιάς που είναι οι γλώσσες στην Ευρώπη, δεδομένου αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Για την φυσική επίσης βιοπικιλότητα, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα κάνει σημαντικές πολιτικές για τη διασφάλιση τους. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτό το ζωντανό πολιτιστικό κληροδότημα που έχουμε, που είναι σημαντικό και έχει και διάφορα ατού, κυρίως για διάφορες ε, διασυνοριακές περιοχές όπου η δυνατότητα κατανόησης των μεν, των δε, ένθεν και ένθεν των συνόρων είναι και θέμα κατανόησης περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, όπως ξέρουμε, τις 23 ε, επίσημες γλώσσες, αλλά δεν επωφελείται μόνο από τις επίσημες γλώσσες. Από τη στιγμή που υπάρχει μία γλωσσική κοινότητα που χρησιμοποιεί μία άλλη γλώσσα, και αυτή αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και πρέπει να την ε, μεταχειριζόμαστε ίσης όρις με τις άλλες. Υπάρχουν βεβαίως κάποιες οι οποίες απειλούνται και εδώ θα πρέπει να επαγρυπνούμε και να αναλάβουν δεσμεύσεις τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να είναι πιο δυναμικά υπέρ την προστασία τους. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Την διγλωσία εκγενετής, δηλαδή από τις πρώτες μέρες της γέννησής του το παιδί να μπορεί να μαθαίνει και να κατέχει σιγά σιγά δύο γλώσσες. Όχι μόνο για τις απειλούμενες, αλλά για όλες. Όλοι οι νέοι Ευρωπαίοι θα πρέπει ευθύ εξ αρχής να μπορούν να είναι δίγλωσσα. Διότι από τη στιγμή που γίνεται κάτι τέτοιο, καταρχήν αναπτύσσει κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών τη δυνατότητα να μάθει μια τρίτη, μια τέταρτη και να συνεχίσει. Κάτι άλλο το οποίο θα επίση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι το γεγονό ότι στα δύο τελευταία ε, πολιετή δημοσιονομικά προγράμματα δόθηκαν διάφορες ενισχύσεις υπέρ των γλωσσών, κυρίως των πλέον αδύναμων και απειλούμενων, αλλά δεν είναι αρκετή. Τι προτείνει η εκθεσή μου. Να κινητοποιήσουμε εκ νέου τα κράτη-μέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να υποστηρίξουν τις πολιτικές διασφάλισης αυτών των γλωσσών οι οποίες υπάρχουν στα πλαίσια των κοινοτήτων των οποίων οι γλώσσες απειλούνται. Με ποια μέσα. Με όλα τα μέσα τα Δεν υπάρχει πρόγραμμα σήμερα που να μην μπορεί να προσαρμοστεί με τρόπο που να βοηθήσει αυτό τον εγκάσιο στόχο μέσω των ε, κοινοτικών ταμείων, μέσω των κονδυλίων που προβλέπεται την ενίσχυση της εκπαίδευσης κτλ. Επίσης, ένα πρόγραμμα που θα μας επιτρέψει από την ε, πολύ νέα ηλικία στα παιδιά να έχουν δύο μητρικές γλώσσες είναι πρωταρχική σημασία ώστε να μπορέσει να υπάρχει ευκολία στην μετάδοση αυτών των γλωσσικών γνώσεων τη μια γενιά στην άλλη. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε τι μπορεί ε, να, κάνουν αυτές οι κοινότητες οι οποίες δεν είναι και τόσο πολυάριθμες που μιλούν μια τέτοια ε, γλώσσα. Θα πρέπει αυτό το κριτήριο ε, να το λάβουμε υπόψη ώστε σε αυτές τις αδύναμες γλωσσικά όπως λέμε και αεροκατοικημένες περιοχές να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Να υποστηρίξουμε προγράμματα, προγράμματα ποικιλόμορφα ε, μακροπρόθεσμα που αφορούν πάρα πολλά θέματα, τα μίντια, την καθημερινή ζωή, όλα τα μέσα, την εκπαίδευση και τέτοιους προγράμματα να τα υποστηρίξουμε. Ώστε οι γλωσσικά δύναμες αυτές κοινότητες να εμπλωτιστούν, να αποτελέσουν δίκτυα σε επίπεδο κρατών ή περιοχών υπάρχουν τέτοιου είδους δίκτυα, σε επίπεδο μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, και υπάρχουν και διάφορες πρωτοβουλίες υπέρ των απειλούμενων ε, γλωσσών. Εγώ ως ε, ε Γάλλος που κατάγεται από την Κορσική, έχω παραστεί σε διάφορα φεστιβάλ τραγουδιού για τις μειονοτικές αυτές γλώσσες. Και στις προσπάθειες, έχω δει τις προσπάθειες που καταβάλλονται να ενισχυθούν οι γλώσσες αυτές. Θα πρέπει επίσης να συνεχίσει η UNESCO την εργασία της και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουμε και κάποια ενίσχυση σε αυτά τα προγράμματα. Τελειώνοντας την παρουσίασή μου, θα ήθελα να πω ότι για μας είναι σημαντικό να προστατεύσουμε, να ενισχύσουμε αυτές τις κοινότητες, να διασφαλίσουμε ε, το τι έχει επιτευχθεί μέσα σήμερα, τα κεκτημένα. Υπάρχει μια ιστοσελίδα, η Αντομίνφο, για, που παρέχει ενημέρωση σχετικά με τα κοινοτικά προγράμματα και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες οι γλώσσες να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, Europe Creative και να μην αποκλειστεί καμία περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα που ομιλείται στα κράτη-μέλη. Διότι όλες αυτές οι γλώσσες είναι μέρος της πολιτιστικής ζωντανής κληρονομιάς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε. Äh, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλω να επισημάνω σε όλους ότι ε, θα πρέπει να διαβάσετε και την ε, έκθεση της Επιτροπής ε, Πολιτισμού στη Λαπωνία και θα δείτε τι σημαίνει απειλούμενες γλώσσες. Είμαστε σε μία πόλη στο Ίνερε και εκεί υπάρχει μόνο μία γλώσσα, το Σάμι, που την μιλάνε 380 άνθρωποι. Και οι κάτοικοι αυτής της περιοχής επιθυμούν να διατηρήσουν τη γλώσσα τους. Αυτοί λοιπόν έχουν παιδικούς σταθμούς όπου τα παιδιά τους από πολύ μικρή ηλικία ακούν μόνο αυτή τη γλώσσα. Μεγαλώνουν με αυτή την ηλικία, ε, με αυτή τη γλώσσα και τη φέρνουν στο σπίτι τους. Δηλαδή από τα παιδιά έρχεται η ε, γλώσσα στα σπίτια Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, γιατί νομίζω ότι πρόκειται για μια θαυμάσια γλωσσική πολυμορφία που έχουμε. Εμείς το ζήσαμε στο πετσί μας και πραγματικά συγκινηθήκαμε και θέλω να σας πω ότι σήμερα τα θυμήθηκα όλα αυτά και ελπίζω με το κείμενο που έχουμε καταρτήσει θα ασχοληθούμε επί της ουσίας με τις ε, απειλούμενες γλώσσες. Απειλούμενες γλώσσες είναι αυτές που δεν μιλούνται σχεδόν καθόλου και είναι όμως αναπόσπαστο κομμάτι και του παρόντος αλλά και του παρελθόντος μας. Ο κύριος Τάκουλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ συγγνώμη πρέπει να φύγω να πάω σε μια άλλη επιτροπή. Έχουμε ένα πρόβλημα εμεί εδώ γιατί έχουμε πολλέ συνεδριάσει επιτροπών ε, παράλληλα και πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μα να εξασφαλίσουμε το γεγονός ε, ότι η γλώσσα Σάμι αλλά και άλλες ε, απειλούμενες με εξαφάνιση γλώσσες να λάβουν την προστασία που χρειάζονται ώστε να μπορούν να αναβιώσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν και τον κύριο Αλφόνση για την εξαιρετική του έκθεση. Σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ικανοποιημένος με το κείμενο λαμβάνει υπόψη όλες τις μικρότερες και παπιλούμενες γλώσσες και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερος. Όπως είπε και η πρόεδρος, Όταν πήγαμε στη Βόρεια Φινλανδία, είδαμε ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτό που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη L και στην παράγραφο 1. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι η οικονομική βοήθεια για την προστασία των μειονοτικών γλωσσών έχει μειωθεί σημαντικά και αυτό δεν είναι ε, σωστό. Πρέπει να προστατεύσουμε το μέλλον των γλωσσών αυτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο και όπως είπε άλλωστε και η πρόεδρος, ε, αυτά τα γλωσσικά προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται και στη Φινλανδία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιες μειονοτικές γλώσσες είναι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, τις οποίες πρέπει να υποστηρίξουμε. Επικροτώ λοιπόν την έκθεση του κυρίου Αλφόνση και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε σε αυτήν την οδό που μας έδειξε ο κύριος Αλφόνση. Συγγνώμη που πρέπει να φύγω. Και εγώ, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Αλφόνση για τη δουλειά του, για ένα θέμα ε, για το οποίο ε, νιώθω ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί εγώ προέρχομαι από μια τέτοια περιφέρεια. Ε, κάθε φορά πρέπει να γίνεται μια προσπάθεια προστασία, προστασία των γλωσσών. Για μένα είναι τα καταλανικά, για τον κύριο Αλφόνση είναι τα κορσικανικά. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να φέρουμε πιο κοντά και τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει να υπάρχει μια πολιτική για τη δέσμευση της Ευρώπης, για την διάσωση της πολιτιστικής και γλωσσικής κληρονομιάς μας και πρέπει να, ε, να ευαισθητοποιήσουμε εκ νέου ε, τον κόσμο γιατί πρέπει να προστατεύσουμε αυτή τη γλωσσική ποικιλομορφία. Ο Φρανσουά Αλφόνση το είπε, αλλά θα ήθελα να το πω και εγώ. Μια γλώσσα είναι μια κληρονομιά μια κοινότητα, αλλά και ολόκληρη τη Ευρώπη. Και δεν μπορούμε εμεί ω Ευρωβουλευτέ ε, να βλέπουμε ότι υπάρχει ε, διάβρωση τη γλωσσική ποικιλομορφία και να το επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι και γι' αυτό ακριβώ υποστηρίζω όλα αυτά που είπε ο συνάδελφο στην εκθεσή τη, όχι μόνο μόνο εκ μέρους της Επιτροπής αυτής, αλλά και ε, είναι και προσωπική μου άποψη. Ε, τα καταλανικά, 8 εκατομμύρια πολίτες το μιλούν και παρά το γεγονός ότι λέμε ότι είναι επαπειλούμενοι, υπάρχει πραγματικά μια κοινότητα που ενδιαφέρεται για αυτές τις γλώσσες, ενδιαφέρονται όμως και όλες οι Ευρώπης. Ε, δεν, δεν υπάρχει, ας πούμε, μια ε, καμπίνα μετάφρασης γλώσσας αυτής. Πρέπει όμως να την προστατεύσουμε. Ξέρετε ότι υπάρχει εκπαίδευση στη γλώσσα αυτή και χαίρομαι πάρα πολύ ε, που ακούω ότι υπάρχουν βρεφονιπιακοί σταθμοί από από πολύ μικρή ηλικία, εξ ήχων αρχίζουμε να μιλάμε μία ε, ε, δεύτερη γλώσσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τότε είναι σαν σφουγγάρια τα παιδιά και τότε αρχίζουν πραγματικά να μαθαίνουν γλώσσε. τότε είναι πιο εύκολο να μάθουν πιο πολλέ γλώσσε. Γι' αυτό πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, κινητοποιήσει όλου του τους σπόρους για να βοηθήσει την κατάσταση αυτή, να βοηθήσει τι τοπικέ και περιφερειακές αρχέ, να ασχοληθούν και να ανησυχήσουν για αυτέ τι επαπειλούμενες γλώσσε, γιατί σημαίνουν πολλά πράγματα για αυτού που τι μιλούν. Είναι σημαντικό τμήμα τη κληρονομιά μα. Υπάρχει και η πολιτιστική μας ε, διαφορά, την οποία θέλουμε πραγματικά να την υποστηρίξουμε, ειδικότερα σε μια περίοδο αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης. Αυτές οι λιγότερο χρησιμοποιημένες γλώσσες πρέπει πραγματικά να τύχουν υποστήριξης. Είναι ένας πλούτος πολιτιστικός, αλλά είναι και πραγματικά μια ευκαιρία για την Ευρώπη να προσεγγίσει τους πολίτες της. Έχει η Ευρώπη ένα ρόλο μακροπρόθεσμα ε, να διαδραματίσει για τη διατήρηση αυτής ακριβώς πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν πεθαίνει όμως η γλώσσα η καταλανική, ε, σας το λέω για να το γνωρίζετε. Μιλάμε για επαπειλούμενε γλώσσε τώρα, έτσι, το επενθυμίζω αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μακλάρκεν έχει το λόγο. Thank you, chairman. Um, Ευχαριστώ πολύ η συνάδελφο, την οποία εκπροσωπώ δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα για να συζητήσει αυτό. Είναι στον τριμερή διάλογο τη Επιτροπή ΕΚΟΝ, αλλά χαίρεται όλος ιδιαίτερος ε, που υποστηρίζει την ε, έκθεση ε, της, του κυρίου Αλφόνση. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που θέλει να τονίσει ιδιαίτερα, την ευθύνη μα για τη, για τη διατήρηση των γλωσσών αυτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη τη γλωσσική ποικιλομορφία στο παρελθόν, αλλά όπω λέει και η έκθεση, πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία για στι επαπειλούμενε γλώσσες, γλώσσες που χρειάζονται υποστήριξη. Ακούσαμε πολύ ανησυχητικέ ε, στατιστικές για τον ανησυχητικό βαθμό στον οποίο γίνονται κάποιε γλώσσε επαπιλούμενες και μιλάω για την Ουαλία για παράδειγμα. Ε, η γλώσσα αυτή στην Ουαλία εξακολουθεί να ε, ομιλείται περήφανα όμως ε, είναι η μικρότερος ο αριθμός ε, των ε, ανθρώπων που τη μιλούν. Είναι κρίμα που επικεντρωνόμαστε μόνο στις επαπειλούμενες γλώσσες, γιατί και η ουαλική γλώσσα είναι μία γλώσσα η οποία θεωρούμε ότι πραγματικά ε, αντιμετωπίζει πρόβλημα. Έχει όμως ε, τύχη υποστήριξης και γι' αυτό έχει αναβιώσει. Είναι λοιπόν ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης με την προώθηση δραστηριοτήτων υπέρ των γλωσσών αυτών. Η ψηφιακή τεχνολογία επίσης, ε, τα κοινωνικά μίντια, facebook, twitter, ε, μπορούν να δώσουν ε, μεγαλύτερη όθηση στις επαπειλούμενες γλώσσες. Πρέπει να υποστηρίξουμε και τη γλωσσική, τη γλωσσική κοινότητα ότι στην προσπάθειά τους να δράξουν ευκαιρίε για να ε, προωθήσουν τις γλώσσες τους. Πρέπει επίσης ε, να υπάρξουν πρωτοβουλίε σχετικά με αυτό ε, και είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να υποστηρίξουμε σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής τις επαπειλούμενες γλώσσες πρέπει να υποστηρίξουμε ε, την άνετη χρήση των ε, γλωσσών αυτών ε, στον επαγγελματικό χώρο και ε, στο σπίτι τους, γιατί πραγματικά με αυτόν τον τρόπο μπορεί μία γλώσσα να τη μεταλαμπαδεύσει η μία γενιά στην άλλη. Ευχαριστώ πολύ. Χέλγα. Ευχαριστώ θα ήθελα να επανέλθω στην ε, επίσκεψη της αντιπροσωπεία μας ε, στην περιοχή των Σάμι στη Λαπωνία. Ήταν πραγματικά μια πολύ συγκινητική επίσκεψη. Εμένα με συγκίνησαν αυτοί οι καταπληκτικοί άνθρωποι που θέλουν τόσο πολύ να βοηθήσουν τη μειονοτική τους γλώσσα. Και υπάρχουν και δύο ακόμη γλώσσες ε, Σάμι, τα βόρεια Σάμι και τα σκόλτ Σάμι δεν το ήξερα αυτό στο παρελθόν. Πρέπει να το ομολογήσω ότι υπάρχουν, τόσο, ότι υπάρχουν τόσες γλώσσες στον Σάμι και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα να δω ότι ήταν πραγματικά τόσο φωσιωμένοι στην κατανόηση της γλωσσικής και πολιτιστικής επικοινωνία και ότι με τη δική μας υποστήριξη, με ευρωπαϊκά κονδύλια, όχι μόνο με εθνικά κονδύλια, πραγματικά οικοδόμησαν μια ολόκληρη προσπάθεια ευρεπονιπηρικού σταθμού, σχολεία για να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς ε, και μέσω αυτού του τρόπου επιστρέφει αυτή η δυνατότητα στις οικογένειες ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν. Είναι οι μόνοι αυτόχθονες ε, ε, της, ε, Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίσουμε αυτό και είναι πάρα πολύ αφοσιωμένοι στις αξίες τους, στη γλώσσα τους. Δεν είναι εχθρικοί στα φιλανδικά, προς τα φιλανδικά. Υπάρχει μια έννοια συνύπαρξης. Εκείνοι επενδύουν στο δικό τους πολιτισμό και παράλληλα βέβαια μιλούν και φιλανδικά και ζουν στη Φιλανδία. Αλλά ε, κατά την άποψή μου, όταν ήμουν εκεί, αυτό που ένιωσα είναι ότι είναι ένα πολύ καλό και πλούσιο συνδυασμό. Έχει τη δική σου μειονωτική γλώσσα, όμω, είσαι τμήμα της ε, του φιλανδικού πολιτισμού επίση, Δεν είναι κανένα επιθετικό ούτε εχθρικό προ τα φιλανδικά. Υπάρχει ένα πολύ καλό συνδυασμό, μια συνύπαρξη. Και γι' αυτό ελπίζω ότι αυτό θα είναι τμήμα και τη δική μα προσέγγιση όταν θα θελήσουμε να καταπολεμήσουμε την απειλή κατά των γλωσσών αυτών. Θέλουμε να αναβιώσουν αυτές οι γλώσσες, αλλά από την άλλη δεν θέλουμε να είναι ένας ένας, μια σκληρή μάχη ε, με άλλους πολιτισμούς. Ε, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτήν την εμπειρία που είχαμε με τους Σάμι όταν θα πρέπει να μεταγράψουμε την ε, πολιτική μας. Κυρία Παλιαδέλη. παρατήρηση της Χέλγα γιατί πραγματικά είναι πιθανό πρώτον γλώσσες που δεν είναι σε κίνδυνο να θεωρηθούν ότι είναι σε κίνδυνο παρόλο που μιλούνται από μεγάλους αριθμούς να εκτιμώνται ότι είναι σε κίνδυνο από μεγάλους αριθμούς ε, πληθυσμών να έχουν γραπτή μορφή ή να χρησιμοποιηθούν για ε, ε, επιδιώξεις που δεν σχετίζονται άμεσα με τον πολιτισμό. Καταρχήν να πω ότι για την δική μου εκτίμηση οι άμεσα επαπειλούμενες γλώσσες με εξαφάνιση είναι οι γλώσσες που μεταδίδονται προφορικά. Οι γλώσσες που έχουν γραπτή μορφή, τα κείμενά τους μεταφράζονται, μπορούν να μελετηθούν, είναι μια άλλη ιστορία. Καταρχήν λοιπόν θα πρέπει να δούμε και αυτή την ενότητα που είναι οι προφορικές γλώσσες και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι επομένως είναι κατά κύριο λόγο επαπειλούμενες. Από αυτή την άποψη οι κοινότητες Σάμι δίνουν και ένα άλλο ενδεχόμενο στοιχείο το ότι συνεργάστηκαν με ένα πρόγραμμα Interreg οι δύο χώρες, η Φιλανδία και η Νορβηγία για την υποστήριξη αυτής της, ε, αυτών των διαλέκτων. Απ' την άλλη μεριά θεωρώ ότι ε, πρέπει να διασφαλίσουμε τον όρο επαπειλούμενη σε διαφοροποίηση από το minority ή regional γιατί ο στόχος μας είναι να σώσουμε την πολιτική κληρονομιά της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το γλωσσικό πεδίο. Όχι να δημιουργήσουμε αφορμές για άλλου είδους διεκδικήσεις που ίσα ίσα θα μποϊκόταραν, θα δημιούργησαν ζητήματα σε τέτοιου είδους προθέσεις όπως είναι η πολιτιστική, ε, η διατήρηση της πολιτικής κληρονομιάς. Ως ε, shadow ε, ως ε, στο κείμενο του κ. Αλφόνση, τον οποίο ευχαριστώ πολύ, ε, ε, δηλώνουν ότι δεν υπάρχει ούτε μία φορά η χρήση του όρου minority ή regional language όπως άλλωστε πρέπει να είναι σε αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση και ότι πιστεύω ότι πρέπει να τονιστεί, θα το προτείνω με τις τροπολογίες μου, η, η θέση της ε, Επιτροπής Πολιτισμού με κύριο στόχο να προστατέψει την πολιτιστική κληρονομιά όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις γλώσσες. Όχι να δώσει διεξόδους σε άλλες επιδιώξεις που υπερβαίνουν και, τους, και τις προθέσεις μας και, είναι, και ίσα ίσα αντιβαίνουν και στην ε, ε, ευρωπαϊκή ιδέα και στην ενότητά της. Επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, θα το προτείνω σε ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ τον κύριο Αλφόνση έτσι κι αλλιώς. Vielen Dank. Herr Κύριε Τούκης. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ελφόνζη. Νομίζω ότι ο Κορσικανός ε, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος ε, για να βρίσκεται στη θέση του εισηγητή αυτής της έκθεσης. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής για την έκθεση αυτή. Και μπορώ να σας πω, επειδή και εγώ είμαι τμήμα μειονότητας ε, στην ε, Ρουμανία, κυρία Παλιαδέλη, το θέμα της μειονότητα των μειωτικών γλωσσών δεν μπορεί κανείς να το αποκόψει από τις επαπειλούμενες γλώσσες ε, και το πρόβλημά τους. Βεβαίως πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο γλωσσικό πρόβλημα. Αυτό πρέπει να τονίσουμε, αλλά μπορώ να σας πω ότι πριν από 90 χρόνια 45% της Τρανσιλβανίας μιλούσαν γερμανικά, ουγγρικά και άλλες μειονοτικές γλώσσες και τώρα έχει μείνει 20% της παλιάς Τρανσιλβανίας που χρησιμοποιεί την ουγγρική γλώσσα. Βεβαίως υπάρχουν ε, γλώσσες στην Ευρώπη που πραγματικά εξαφανίζονται και άλλες που εν μέρη απειλούνται με εξαφάνιση. Ας πούμε δύο τρίτα της, ε, στα δύο τρίτα της Τρανσιλβανίας ε, τα ουγγρικά ή τα γερμανικά εξαφανίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά στο Ζίμπενμπουργεν. Πρέπει να τονίσω λοιπόν ότι το πρόβλημα των επαπειλουμένων γλωσσών δεν είναι μόνο γλωσσικό και πολιτιστικό, αλλά είναι και θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικό ζήτημα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η βλάχη της Σερβίας. Η Σερβία τώρα είναι υπό ένταξη χώρα. Στην κοιλάδα Τιμόκ, ε, σε 12 σχολεία, η ρουμανική γλώσσα των βλάχων εισήχθη υπό την πίεση της Ρουμανίας, η ρουμανική κυβέρνηση και του Προέδρου Πασέσκου. Υπάρχει άλλη μια κοινότητα στη Ρουμανία, η Τσάγκου Ούγρι, τον οποιων η γλώσσα, που είναι μια διάλεκτος της Ουγγαρίας, σχεδόν εξαφανίζεται. Ή γνωρίζουμε, ας πούμε, ε, του, ε, τα δικαιώματα των Σάμι. Η γνωρίζετε ότι η κοινότητα των Σάμι έχει μια περίπλοκη αυτονομία, εξασφαλίζονται τα δικαιώματά τους, τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και τα δικαιώματά τους ως μειονότητας. Η Γαλλία, για παράδειγμα, δεν υπέγραψε την χάρτα ε, περιφερειακών ε, και μειονοτικών ε, δικαιωμάτων. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες διαφορές, αυτό θέλω να πω, και πρέπει να τονίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ε, πολιτικά ε, δικαιώματα ε, και τα γλωσσικά δικαιώματα είναι συνδεδεμένα και πρέπει να ληφθούν υπόψη με διάφορες τροποποιήσεις στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπόρης. Ευχαριστώ. Πρόκειται για σημαντική έκθεση, διότι πρέπει να τονίσουμε και την πολιτική ε, οπτική γωνία αυτού του προβλήματος των απειλούμενων γλωσσών. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και να το εξετάσουμε περαιπέρω. Οποιαδήποτε ιδέα αφορά τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων με στόχο μελέτες για τις απειλούμενες γλώσσες είναι σωστό και αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια του προγράμματος Creative Europe. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα πανεπιστήμια που συχνά μελετούν τις γλώσσες που απειλούνται στα κράτη-μέλη, αλλά συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης τέτοιου είδους ερευνών και μελετών. Κυρίως και για να μιλήσει κανείς με γυρεότερους ανθρώπους που έχουν πείρα στην ε, ομιλία και στο χειρισμό αυτής της γλώσσας είναι σημαντικό. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά για να βοηθήσουμε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που ασχολούνται με την εκμάθηση και διατήρηση των ευρωπαϊκών γλωστών. Επίσης πιστεύω ότι η υποστήριξη της διδασκαλίας τέτοιου είδους απειλούμενων γλωσσών στα παιδιά έχει να κάνει πολλές φορές και με κάποιες γλωσσικές εθνικές μειονότητες. Το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο δίδει χρήματα για να βελτιώσει την κατάσταση της κατάρτισης των καταρτιστών, εκπαίδευση των, κατα... των εκπαιδευτών. Αυτό είναι σημαντικό για τους δασκάλους για να μπορούν ε, σωστά να διδάσκουν τις γλώσσες αυτές τις απειλούμενες ή άλλα θέματα ε, σε αυτές τις γλώσσες. Θα πρέπει λοιπόν και με την υποστήριξη του Κοινωνικού Ταμείου να παράσουμε βοήθεια. Επίσης, τελικά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι, πρώην, οι χώρες της πρώην κεντρικής ε, ε, Ευρώπης, δηλαδή 12 με 13 γλώσσες, έχουν την εμπειρία μιας πολιτικής που έγινε επί χρόνια, όπου οι μειονοτικές γλώσσες, αν θέλετε, είχαν σβηστεί από το χάρτη. Έγιναν προσπάθειες να σβήσουν από το χάρτη. Και πολλές φορές στην Πολωνία Φελιππίν, στην Νότια Σιλεσία υπάρχουν ε, ε, ε των ΛΕΜ, των ε, Ουκρανών που μετατοπίστηκαν στην Πολωνία για να εξαφανιστούν πολιτιστικά αν θέλετε από την Ουκρανία. Μπόρεσαν όμως να ξανακερδίσουν τη γλώσσα τους ε, οι άνθρωποι εκεί στην Σιλεσία ε, μάζεψαν πάρα πολλές πληροφορίες, κάνουν διάφορα φεστιβάλ, οι νέοι αν θέλετε είναι ενωμένοι μέσω της γλώσσας αυτής της κοινούς, κοινής που μιλούν. Πιστεύω λοιπόν ότι η γλώσσα μπορεί να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους να ξαναιφάνουν αυτό τον ιστό, τον πολιτιστικό που είναι τόσο σημαντικός για τη ζωή τους. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα οικονομικά κονδύλια για να αποτρέψουμε το θάνατο αυτών των γλωσσών που ήταν πλούτος για κάποιους λαούς για αιώνες. Σύστημα ε, ακόμη και στην ε, παγκοσμιοκόμηση των γλωσσικών συστημάτων θα πρέπει περαιτέρω να βοηθήσουμε μια τέτοια κατάσταση. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω ότι και εγώ είμαι ευγνώμων στον συνάδελφο κύριο Αλφόνση για όλα αυτά που μας είπε και βεβαίως και η έκθεση του είναι πάρα πολύ σημαντική. Ομολογώ ότι σκέφτηκα το εξής. Ε, πάρα πολλές ε, από τις γλώσσες που μιλάμε ε, και δεν εξαφανίζονται τώρα πια. Είναι όμως το, η συνέχεια γλωσσών που εξαφανίστηκαν, ας πούμε το, τα λατινικά. Ε, ακόμα και η Εκκλησία σήμερα δεν μιλάει λατινικά. Ο Πάπας όταν μιλάει, μιλάει ισπανικά, ιταλικά. Δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό, ότι προφανώς υπάρχει ας πούμε αυτή η ιστορική εξέλιξη και εμείς δεν μπορούμε να την απαρνηθούμε. Ε, το θέμα των ε, πανεπιστημίων νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό από την επιβίωση. Οι Σάμι καλούνται να επιδιώσουν τον άλλον ε, που ε, θέλουν να τους κατακτήσουν. Ε, το ίδιο συνέβη και με τα λατινικά που επικράτησαν γιατί ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Άρα δηλαδή με τις γλώσσες τι γίνεται, προχωράμε και με το πολιτικό γίγνεσθε. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μην τις χάσουμε τις γλώσσες αυτές ως πολιτιστική κληρονομιά. Άρα δηλαδή είναι σημαντικό να υπάρχουν οι πανεπιστημιακές σχολές. Εγώ ας πούμε στην Ιταλία είδα στην, ε, σε ένα τμήμα, σε μια έδρα γλωσσολογίας, ε, χάνονται όλο και περισσότερο κάποιες γλώσσες γιατί δεν είχαμε λεφτά να τις ε, χρηματοδοτήσουμε. Εγώ, α πούμε, υπεραμείνθηκα στη δική μου τη σχολή των Ουγγρικών μέχρι θανάτου. Βεβαίω κάποια στιγμή και εγώ δεν μπορούσα να συνεχίσω. Τι θέλω να πω με άλλα λόγια. Ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε στην έκθεση ότι πρέπει να υπάρχει η επιβίωση κάποιων ε, κοινοτήτων ε, που μιλάνε ε, μια γλώσσα, να υπάρχουν Τη παιδική σταθμή. Αλλά εντάξει, το πανεπιστήμιο, εγώ επιμένω, το πανεπιστήμιο είναι ο βασικός φορέας διαφύλαξης των γλωσσών. Εντάξει, καλέ και καλή και η παιδική σταθμή δεν είναι το ίδιο. Ε, και εν πάση περιπτώσει, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποιες τοπικές γλώσσες, αυτή μεταξύ τη Πιεμόντε και τη Γαλλία, ε, όπου σε αυτή τη γλώσσα υπάρχουν έγγραφα πάρα πολύ σημαντικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ε, απόκτηση στοιχείων. Σίγουρα δεν πρέπει να χαθούν όλα αυτά που υπάρχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, όμως, λέει πρόεδρος, ε, δεν φαντάζομαι ότι πιστεύει ότι θα χαθούν τα ογκρικά επειδή δεν διδάσκονται πια στην Ιταλία. Ε, γιατί το να το λέτε αυτό κάπως ξεφεύγουν το θέμα. Όχι, εντάξει. Η Σαμπίνε. Και εγώ θέλω να πω το εξή. Νομίζω ομιλώ και εξάλλον λέγοντας ότι δεν πρέπει όλα τα προβλήματα του κόσμου να τα λύσουμε με αυτή την έκθεση. Ε, πρέπει λοιπόν να προσέξουμε λιγάκι, να εστιάσουμε την προσοχή μας σε γλώσσες που πραγματικά απειλούνται να εξαφανιστούν πλήρως. Ας πούμε, η γερμανική μειονότητα στο Βέλγιο. 380.000 είναι. Ε, βέβαια, εντάξει, έχουν μειωθεί τώρα, έχουν πάει στου 97.000 ε, και έχουν μητρική γλώσσα γερμανικά. Ε, Κανεί όμω δεν λέει ότι απειλούνται τα γερμανικά να εξαφανιστούν, γιατί υπάρχουν 90 ή 100 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν μητρική γλώσσα τα γερμανικά. Τι θέλω να πω, να διαφοροποιήσουμε λιγάκι την κατάσταση. Άλλο το Σάμι, το οποίο με πάση περιπτώσει μιλιέται μόνο από 350 ανθρώπου ή αν πρόκειται για μια γλώσσα η οποία ομιλείται από μια μειονότητα μια χώρα, δεν απειλείται όμως με εξαφάνιση, άλλο το άλλο τ' άλλο. Η δεύτερη δεν απειλείται, δεν είναι επαπειλούμενη Απλά και τι άλλο θέμα, να σεβόμαστε την γλωσσική ποικιλομορφία και πέρα από τη μητρική γλώσσα, αυτά να τα πούμε στην έκθεση. Επίσης, να επισημάνουμε στην έκθεση τα προβλήματα που έχουμε, τα οικονομικά, ε, να τα επισημάνουμε όσον αφορά την γλωσσική υποστήριξη και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στη στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Γιατί η δυνατότητα να μεγαλώνει κανεί ε, με δύο γλώσσε, όπω στη Φινλανδία, από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά μαθαίνουν μία γλώσσα ε, στην καθημερινή τους ε, ζωή μέσα από αυτούς τους ε, γλωσσικούς παιδικούς σταθμούς, ε, language and nests όπως τα αποκαλέσαμε. Αυτό είναι ένας πάρα πολύ καλός δρόμος. Αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε και εμείς ε, παραδείγματα, βέλτιστες πρακτικές, παραδείγματα προς μίμηση. Θεωρώ λοιπόν ότι το πολιτικό στοιχείο που κρύβεται πίσω από τη γλωσσική αυτονομία ή πίσω από το δικαίωμα να χρησιμοποιεί κανείς μία γλώσσα στην καθημερινή του ζωή και να τη χρησιμοποιεί ως επίσημη γλώσσα, αυτό να το ξεχωρίσουμε από αυτό που παίζει ρόλο στην έκθεσή μας. Τι παίζει ρόλο? Το να διαφυλάξουμε γλωσσικά την πολυμορφία. Και δεν το λέμε αυτό, ας πούμε, και με τα ζώα ότι όταν ας πούμε απειλείται ένα ζώο από εξαφάνιση δεν λέμε αυτό το είδος ζώου να εισαχθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, το ίδιο ισχύει και για τα ουγγρικά. Δεν μπορεί ας πούμε, να πούμε ότι επειδή τα ουγγρικά απειλούνται από εξαφάνιση να εισαχθούν σε όλες τις γλώσσες και να εντάσσονται παντού. Καταλήν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, εγώ αν δεν γίνει αυτό που σας είπα με τα πανεπιστήμια θα δείτε πώς θα εξελιχθούμε. Ε, Ευχαριστώ την εισηγήτρια για αυτή την πρωτοβουλία, διότι είναι η έκθεση αυτή την κατάλληλη στιγμή. Διότι είναι σημαντικό να πούμε ότι πολύ λίγα κονδύλια γίνονται για την ε, ε κουλτούρα και τη γλώσσα. Πιστεύω όμως ότι η κουλτούρα, η γλώσσα, ε, αυτός ο πλούτος μπορεί να μας οδηγήσει ως Ευρώπη να βγούμε από την κρίση. Θα πρέπει λοιπόν στα πλαίσια του πολιετούς χρηματοδοτικού να κάνουμε κάτι. Δεν πρόκειται μόνο για το σχολείο το επίσημο, για την κατάρτιση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια ώστε να επενδύσουμε στις αξίες τις οποίες αν παραγνωρίσουμε θα χαθούν. Δεν αρκεί για μένα να μιλούμε μόνο για απειλούμενες γλώσσες. Θα πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να τις αναζωογονήσουμε. Όταν κανένας πλέον δεν μιλάει μια γλώσσα, όταν τα παιδιά δεν πηγαίνουν να κάνουν μαθήματα σε αυτή τη γλώσσα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Χάνεται σιγά σιγά η γλώσσα. Στην έκθεση λοιπόν αυτή που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, μιλούμε για προστασία των μειονοτήτων. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις της UNESCO για το θέμα αυτό. Και τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι μειονότητες είναι σημαντικά. Και πρόκειται για κάτι το οποίο έχει, έχει ήδη συζητηθεί. Βεβαίως, οι γλώσσες των μειονοτήτων αποτελούν μία μεγάλη εστία πλούτου. Δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω στον εισηγητή ότι θα πρέπει πραγματικά να ασχοληθεί κατεξοχήν με τις γλώσσες που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Εγώ συμφωνώ εν μέρη με την κυρία Βερχόιεν. Εάν οι αρκούδες από την ε, ε, Ισπανία εξαφανιστούν, αλλά οι αρκούδες της Ρουμανίας δεν εξαφανιστούν, για μένα είναι απώλεια. Οι βλάχοι της ε, Σερβίας και η εκείνη της Τρανσιλβανίας πρέπει εξίσου να μπορέσουν ως κοινότητες να διαφυλαχτούν. Διότι όταν εξαφανίζεται ένα, ένας, εξαφανίζεται και ο άλλος. Όλες τι περιφερειακές μενοτικέ γλώσσες θα πρέπει να τις προστατεύσουμε. Και εγώ πιστεύω ότι η έκθεση του κυρίου Αλφόνση θα δείξει αυτό το θέμα γιατί νομίζω ότι όλοι τελικά θέλουμε όπου ζουν οι άνθρωποι να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους. Αλλά δεν είναι αυτό το βασικό θέμα της έκθεσης. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι οι τροπολογίες αφορούν, ε, θα πρέπει να αφορούν τις επαπειλούμενες γλώσσες. Βλέποντας ας πούμε 50 τροπολογίες για γλώσσες ε, μειονοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ αυτές δεν τις δεχτώ, θα τις απορρίψω. Η έκθεση έχει συγκεκριμένη επικεφαλίδα και πρέπει να γίνει σεβαστή αυτή. Βεβαίω, ε, όποιο δεν με ακούει τώρα, ο κύριος Αλφονσί μετά ε, θα αναγκαστεί να απορρίψει τις ε, τροπολογίες. Το κύριος ε, Τούκης δεν πρόσεχε. Λοιπόν, οι τροπολογίες θα πρέπει να έχουν σχέση με τις επαπειλούμενες γλώσσες και δεν μπορούμε να πάρουμε 30-40 τροπολογίες όπου θα πρόκειται για μία μεγάλη γλώσσα ε, σε μια χώρα. Εντάξει, θα το πει κάπου ο κύριος Αλφονσί, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό θέμα. Η επικεφαλή της έκθεσης είναι διαφορετική. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία από την Κομισιόν. Η κυρία Περέρα σωστά τα λέω. Παρακαλώ. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Αλφόνση για την εργασία του και διότι ασχολείται με το θέμα αυτό Εκτός μικροφώνου, δυστυχώς η πρόεδρος. Δεν ακούμε τι λέει. Παρακαλώ το μικρόφωνο στην πρόεδρο, να μπορούμε να μεταφράσουμε. Λυπάμαι πολύ, δεν ακούμε τι λέει η πρόεδρος. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή κύριο Αλφονσί, ο οποίος ασχολείται με το θέμα αυτό των απειλούμενων με εξαφάνιση γλωστών. Η προσέγγιση για την ε, προώθηση της εκμάθησης ε, των γλωσσών αυτών σε πολύ νεαρή ηλικία είναι κάτι σωστό. Αν τα παιδιά δεν μάθουν αυτές τις απειλούμε με εξαφάνιση γλώσσες, ίσως κάποια στιγμή θα εξαφανιστούν. Οι προσπάθειες λοιπόν πρέπει να επικεντρωθούν εκεί κατά πρώτο λόγο. Δυστυχώς υπάρχουν δυσκολίες στον τομέα αυτό, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί ε, περιορισμένες αρμοδιότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης εμπίπτει στα κράτη-μέλη, σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Και δύσκολα η Κομισιό μπορεί να ενεργήσει με τρόπο πιο δυναμικό και να παρέμβει περισσότερο. Τούτου λεχθέντος. Πρέπει να πω ότι εδώ γίνονται κάποιες επισημάσεις στην Επιτροπή, κυρίως σε σχέση με τα μελλοντικά προγράμματα τα οποία θα έπρεπε να εφαρμοστούν. Πιστεύω ότι η Επιτροπή σας, κυρία Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή συμμετέχει πλήρως στην ε, διαπραγμάτευση των μελλοντικών προγραμμάτων και δεν ε, θα ε, πρέπει το θέμα των προγραμμάτων αυτών να το παραγνωρίσουμε για τη σημασία τους. Πιστεύω ότι εδώ κάτι μπορείτε να κάνετε όταν συζητείτε στην διαπραγμάτευση των προγραμμάτων για αυτό το θέμα. Τώρα, δύο στοιχεία τα οποία θα ήθελα από την πρώτη Επιτροπής να τονίσω, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ε, εκπαιδευτικά προγράμματα και τα προγράμματα κατάρτισης για νέους. Το πρόγραμμα έχει έξι αντικειμενικούς στόχους, ένας από τους οποίους αφορά την πρόθεση της εκμάθησης γνωστών και την γλωσσική πολυμορφία. Κατά συνέπεια, υπάρχει χώρος, πιστεύουμε, στο νέο πρόγραμμα να ληφθούν υπόψη κάποιες από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Δύο από τις προτεραιότητες που εντοπίσαμε στην πρώτη της Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος έχει πρώτα απ' όλα σχέση με στρατηγικές ε, εταιρικέ σχέσεις και με στρατηγική υποστήριξη. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη ευελιξία για να μπορέσουν να επιληθούν κάποια προβλήματα. Και τελική μου παρατήρηση αφορά εσάς και την προσπάθειά σας κυρία Πρόεδρε να περιχαρακώσετε με σαφήνεια τον στόχο της έκθεσης αυτής. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι κάπως αμφίσιμη. Μιλούμε για τις μειονοτικές γλώσσες εν γέννη ή για τις απειλούμενες με εξαφάνιση. Θα πρέπει λοιπόν για να υλοποιήσουμε το στόχο μας να είμαστε απόλυτα σαφείς. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βάτιμο για ένα λεπτό παρακαλώ. Κοιτάξτε, με κάθε σεβασμό ε, για το ταξίδι μας στη Λαπωνία θέλω να πω ότι το πρόβλημα που έθεσα εγώ είναι καθοριστική σημασία και για τον εξή λόγο. Ε, προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να επιβιώσουν τεχνητά κάποιες γλώσσες που εξαφανίζονται για ιστορικούς λόγους. Πρέπει απλά να διαφυλάξουμε την κληρονομιά αυτή. Η κληρονομιά είναι σημαντική όταν μιλάμε για τα πανεπιστήμια, για τα ερευνητικά κέντρα. Όλα τα άλλα είναι απλά ε, προσωρινά μέτρα. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εκείνο που έχει σημασία είναι να διαφυλάξουμε τα έγγραφα. Αυτή είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Πρόεδρος, ακριβώς αυτό είναι το θέμα της έκθεσής μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να χαιρετήσω τις αγωγικές σας παρατηρήσεις. Πιστεύω ότι σε αυτό το ε, παράδειγμα των Σαμίρ στην ε, Βιλανδία και η Χέλγα είπατε ποιο είναι το πρωταρχή σημασία θέμα. Όταν κινητοποιούνται η Ευρώπη και τα κράτη-μέλη καταλήγουμε σε μια κατάσταση η οποία όχι μόνο βελτιώνει τη γλωσσική κατάσταση κάποιων κοινοτήτων αλλά δημιουργεί και ένα κάποιο αίσθημα ενθουσιασμού και υπερηφάνεια των ε, κοινοτήτων που αφορά το πρόγραμμα αυτό. Και υπάρχει και η μεγάλη πολιτική σημασία. Δεν υπάρχει έκθεση η οποία να μην έχει και μια πολιτική αποχρώσα διαφορά. Πιστεύω λοιπόν ότι με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αλλάξαμε κάποια πράγματα ιστορικά στην Ευρώπη. Ε, στην ε, Φιλανθία πριν από τον πόλεμο σίγουρα έγιναν ε, μάχες και αγώνες για το γλωσσικό θέμα. Σήμερα με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και με αυτό που κάναμε αλλάξαμε τα πράγματα. Στην συνθήκη της Λισαβόνας η γλωσσική πολυμορφία είναι μία βασική αρχή. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Τώρα, για τις τι γλώσσα, ό,τι και να μιλάει κανείς, ή μία μειονοτική, ή μία απειλούμενη με εξαφάνιση, τον ίδιο πόνο αισθάνεται στην κοινότητα που ζει αν δεν ικανοποιείται πλήρως. Όταν βλέπουμε ε, από την ε, Ευρώπη το πρόβλημα, είναι κάπως ισοσκελισμένα τα πράγματα. Ή κάποιος βλάχος από τη Ρουμανία χάνει τη γλώσσα του, ή κάποιος Ούγγρος ε, για τους Ευρωπαίους είναι το ίδιο κατά κάποιο τρόπο, διότι βλέπουμε σφαιρικά την πολιτιστική γλωσσική κληρονομιά μας να αποδυναμώνεται, να φτωχαίνει και ξέρουμε ότι αν εξαφανιστεί μια γλώσσα κανείς δεν θα μπορέσει να την ξαναφέρει εν ζωή το, ή ούτε καν η εκκλησία μπόρεσε να κάνει κάτι με τα λατινικά ε, οι Σαμί λοιπόν είδατε ότι δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι με τη γλώσσα η κινητοποίηση από κοινού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για την γλωσσική πολυμορφία είναι ο πολιτικός στόχος. Και βεβαίως δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί όπως στην Φινλανδία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αναγνωρίσουμε εμείς στο Κοινοβούλιο και να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε αυτή η βέλτιστη πρακτική της φιλανδικής γλώσσας να εφαρμοστεί και σε άλλους. Εγώ ως Γάλλος με ε, απογοήτευση είδα παρά τις δεσμεύσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να υπογράψει μία διακήρυξη για την προστασία των μειονοτικών γλωσσών, συγγνώμη, να υπαναχωρεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για μας η συζήτηση αυτή θα πρέπει να καταλήξει σε παροχή βοήθειας αυτών που έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Και να ανοίξουμε μία συζήτηση ώστε ο γλωσσικός πολυμορφισμός, ο γλωσσικός πλουραλισμός να γίνει κανόνα στην Ευρώπη. Και εκεί που μπορεί να είναι δεδομένη από το γεγονός ότι κάποια περιοχή, κάποια χώρα μπόρεσε να είναι ο φυσικός απόγονος, αν θέλετε, αυτής της γλώσσας και τη μιλούν όλοι οι γλώσσοι, γλώσσα, έχει καλώς. Εκεί διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ευκολία για όλους τους πολίτες, διότι είναι πολύ απλό να έχουν πρόσβαση στην εκμάθηση όλων των γλωσσών της Ευρώπης. Αυτό είναι ο στόχος της έκθεσης αυτής. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία κατάσταση που για κάποιες γλώσσες είναι κακή. Υπάρχουν μειονοτικές γλώσσες οι οποίες απειλούνται με εξαφάνιση ε, υπάρχουν άλλες οι οποίες θα γλιστρήσουν προς αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν εκ των προτέρων να κάνουμε ό,τι μπορούμε και όπως είπε η συνάδελφος από την ε, Ουαλία πρέπει να γίνουν προσπάθειες και ακόμη περισσότερες. Πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές που θα καλύπτουν πολλές γενναίες. Δεν πρόκειται για κάτι το συγκεκριμένο που αφορά ένα πρόγραμμα και τελείωση. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για να αντιστραφεί η τάση. Κάθε πολίτης λοιπόν ο οποίος παραδοσιακά έχει πρόσβαση σε μια κουλτούρα και σε μια γλώσσα να την μεταφέρει στα παιδιά του και στους απογόνους του. Ευχαριστώ. Dann wollen wir jetzt mal die Diskussion... Πολύ ωραία λέει Πρόεδρο. Ας κλείσουμε τη συζήτηση και θέλω να σα υπενθυμίσω ε, ότι δεν έχουμε πολύ καιρό για την κατάθεση τροπολογιών και το είδαμε αυτό και χτες. Μέχρι ε, τις 25 Απριλίου, τρεις μέρες δηλαδή, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες. Διότι ήδη το Μάιο πρέπει να ψηφίσουμε. 25 λοιπόν Απριλίου, κατάθεση τροπολογιών και νομίζω εδώ και μία εβδομάδα έχετε το κείμενο, τουλάχιστον στα αγγλικά και στα γαλλικά. Κατόπιν τούτου ε, θέλω να καταλάβετε ότι ε, πρέπει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει ε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, διορία 25 Απριλίου και δεν πρόκειται τόσο ε, για το ποιο υποφέρει, αλλά για το ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τις πραγματικά επαπειλούμενες γλώσσες. Και το πρόβλημα είναι το εξής αναφέρθηκε προηγουμένως. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες να ασκήσουμε επιρροή. Βέβαια, μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούμε να βοηθήσουμε. Βοηθήσαμε στην Σουηδία, στη Φινλανδία. Είχαμε προσκαλέσει και τους Λάπονες να έρθουν εδώ έτσι ώστε επειδή και αυτοί τώρα βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πείσουν τους ε, Σουηδούς να τους δώσουν χρήματα για την διαφύλαξη της πολιτικής τους ε, ταυτότητα. Και το κατάφεραν. Νομίζω αυτό συνέβη και στη Φινλανδία. Άρα δηλαδή μπορούμε να ασκήσουμε επιρροή και μπορούμε να παρακαλέσουμε την Κομισιόν στο πλαίσιο των προγραμμάτων να προσφέρει κίνητρα. Τα περισσότερα πρέπει να γίνονται επιτόπου. Αν όμως εμείς ε, δίνουμε την όθηση, ίσως ε, μπορούν ε, και οι πολιτικοί να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την, τις δικές μας προτάσεις. 25 λοιπόν Απριλίου είναι η προθεσμία. Ευχαριστούμε τον κύριο Αλφόνση και τους αδέλφους και πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 11. Εδώ πρόκειται για τον προϋπολογισμό του 2014. Η κυρία Γένσεν. Λοιπόν, ε, τώρα κάτι πρέπει να διαβάσω. Θα το διαβάσω στα αγγλικά. Δεν μπορώ να μεταφράσω στα γερμανικά, δυσκολεύομαι. Pilot projects and preparatory τα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις και στο παρελθόν ε, η Επιτροπή Προπολογισμών έχει ζητήσει όλες τις ιδέες για πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές ε, δράσεις ε, και μετά ζητούμε από την Επιτροπή να σχολιάσει τη βιωσιμότητα, την εφικτότητα αυτών των προγραμμάτων. Η Γραμματεία θα σας στείλει τα απαραίτητα έντυπα που θα συμπληρώσετε ηλεκτρονικώς. Παρακαλούμε να τα στείλετε πίσω ε, μέχρι τις 23 Μαΐου 12 το μεσημέρι στη γραμματεία του, της Επιτροπής μας. Αν έχετε ιδέες, παρακαλώ αποστείλτε ε, αυτήν, ε, αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Ε, όσον αφορά τώρα την τροποποίηση... Συγγνώμη, 23 Μαΐου διορθώνει η Πρόεδρος. 23 Μαΐου. 23 Μαΐου. Ηλεκτρονικά ε, θα πάρετε όλα αυτές τις πληροφορίες και μετά αν θέλετε μπορείτε να τα αλλάξετε. Στη διαδικασία προπολογισμού υποβάλλουμε όχι τροπολογίε στην πρόταση της ε, Επιτροπής, αλλά στη θέση του Συμβουλίου για την πρόταση αυτή. Αλλά αυτό θα το έχουμε στη διάθεσή μας μόνο, μόνο στα τέλη του Ιουλίου. Προτείνω λοιπόν να ακολουθήσουμε και την ίδια διαδικασία που ακολουθήσαμε και πέρυσι για να να, μην ε, χρειαστεί έκτακτη συνεδρίαση τέλη Αυγούστου. Τον Ιούλιο ψηφίζουμε προπαρασκευαστικές δράσεις και πιλωτικά προγράμματα, ε, όπως επίσης και άλλες τροπολογίες που αυξάνουν ή μειώνουν ε, τα νούμερα που προτείνει η Επιτροπή. Οι τροπολογίες για τον προπολογισμό πρέπει να υποβληθούν στα αγγλικά. Δεύτερον, δίνουμε ε, στην εισηγήτρια οριζόντια εντολή να αποκαταστήσει την, την ε, πρόταση της Επιτροπής για όλες τις δημοσιονομικές γραμμές. Ε, αν υπάρχουν περικοπές όπως πέρσι, θα το κάνει αυτό αυτή τη στιγμή, εγκρίνει τη θέση του το Συμβούλιο. Και τρίτο και τελευταίο, εγκρίνουμε την ε, γνώμη, τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών ε, ε, αναφέροντας τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Ε, ο εισηγητής θα υποβάλει το σχέδιο γνωμοδότησης τον Ιούλιο, θα ψηφίσουμε τον Σεπτέμβριο. Μπορούμε να υποβάλουμε τότε τροπολογίες σε όλες τις γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια διαδικασία ε, που πρέπει να την ακολουθήσουμε. Κυρία Γένσεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Πρόεδρε. Θα θυμάστε ότι ψηφίσαμε κατευθυντήριες γραμμές για το προϋπολογισμό του 2014 ε, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου το Μάρτιο και αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ε, έχουν τρεις πτυχές. Πρώτον, ε, προβληματισμός ε, για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Δεν έχουμε νομική βάση, δεν έχουμε πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και προτείναμε η Επιτροπή να ε, υποβάλει μια πρόταση για τον προπολογισμό του 2014 βάσει της πρότασής της για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτή είναι η πρώτη δυσκολία που έχουμε. Και βεβαίως ε, όλες οι κοινοβουλευτικές επιτρομές, ε, επιτροπές ε, δουλεύουν πολύ σκληρά για να θέσουν τις προτεραιότητές τους ώστε το τμήμα του προϋπολογισμού στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ε, πώς θα συνεχίσουμε δεδομένου ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και βέβαια έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Υπήρχε επίσης μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα αυτό των πληρωμών. Ε, βλέπουμε ε, ότι το Συμβούλιο είναι σε άρνηση σε σχέση με τις ε, ανάγκες ε, των, πιστώσεων ε, υποχρεώσεων. Κάνει σαν να μην καταλαβαίνει ότι όταν λαμβάνεις μια υποχρέωση κάποια στιγμή πρέπει να πληρώσεις την υποχρέωση αυτή, για την υποχρέωση αυτή. Κάτι το οποίο έχουμε και εμείς ως πρόβλημα και βέβαια πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πρέπει να το, ζήσουμε, να, το, λύσουμε αυτό το πρόβλημα είναι το θέμα των ε, πολιτικών προτεραιοτήτων όπως ε, η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων που αφορά βέβαια και τη δική σας επιτροπή γιατί αφορά κυρίως την εκπαίδευση ε, το, όπως επίσης και τη στρατηγική 2020. Υπάρχουν όμως και άλλες προτεραιότητες και φυσικά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικές οι προτεραιότητες της Επιτροπής Πολιτισμού. Είδαμε τώρα ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει έναν ε, ενδεικτικό ε, πίνακα που δείχνει ε, τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Φεβρουάριο, στις 7 και 8 Φεβρουαρίου όταν συνεδρίασε. Για τη δική σας Επιτροπή αυξάνονται τα κονδύλια για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά όταν ε, βλέπουμε τις διάφορες κατηγορίες ε, δεν είναι πολύ καλή η μεταχείριση. Ας πούμε το πρόγραμμα για τους πολίτες ε, δεν τα πάει πολύ καλά. Πρέπει να, σημαντικό, να σημόμαστε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι αρχή προϋπολογισμού, δεν ομοθετεί Οπότε μπορείτε βεβαίως να αμφισβητήσετε και να αγωνιστείτε κατά της πρότασης αυτής ε, και πρέπει να το κάνετε και μάλιστα σύντομα να εκφράσετε και τις απόψεις σας ε, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στη διαπραγματευτική ομάδα που θα διαπραγματευτεί τα θέματα αυτά. Εγώ είμαι στη διαπραγματευτική ε, ομάδα, θα ακούσω λοιπόν πολύ προσεκτικά αυτά που θα, που θα πείτε σήμερα αλλά βεβαίως ε, είμαι εδώ για να καλύψω και τις άλλες πτυχές του προπολογισμού 2014 και για να σας ακούσω και γι' αυτό. Είπαμε από πλευράς Κοινοβουλίου ότι η Επιτροπή πρέπει βεβαίως να χρησιμοποιήσει τη, βάση, την πρότασή τη δική της πρόταση ως βάση για ε, τον προϋπολογισμό του 2014, όμως η Επιτροπή είπε ότι έχει προσέξει ότι ε, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, συνεδρίασαν και ότι μπορεί ο προπολογισμό 2014 να συμπεριλάβει κάποιες περικοπές ε, τις οποίες πρότεινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, κατά τα τέλη Μαΐου υποθέτω ότι θα έχουμε μια τέτοια πρόταση και βέβαια ως αυτό προσθέτει στο πρόβλημα που έχουμε με τη διαδικασία του προϋπολογισμού. Αυτά έχω να σας πω ε, για την ώρα. Θα ακούσω τι έχετε να πείτε και ε, βεβαίως θα επανέλθω όταν έχει προχωρήσει η διαδικασία για να εξασφαλίσω ότι βεβαίως ε, συμπεριλαμβάνουμε στη δική σας, τη δική, δικές σας απόψεις στη διαδικασία προπολογισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Γένσεν. Το συζητήσαμε στους συντονιστές αυτή το έγγραφο της Επιτροπής. Στα γερμανικά δηλαδή θα έλεγα ότι θα πρέπει να προσέξουμε όλοι πάρα πολύ και αυτό δεν το κάνουμε. Έχετε πολύ απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι το Συμβούλιο δεν είναι νομοθετικός εταίρος. Έχουμε ένα έγγραφο και συζητάμε για το έγγραφο αυτό. Και εχθές λοιπόν συζητήσαμε γι' αυτό είπαμε ότι είναι απαραίτητο να πούμε στον κύριο Λαμασούρ και στο Συμβούλιο τι ακριβώς επιθυμούμε. Παραδείγματο χάρη, ανεξάρτητα από το ότι η Επιτροπή στον τομέα της παιδείας προσέθεσε κάποια κονδύλια, όχι και πάρα πολλά, αλλά με πάση περιπτώσει είναι σημαντικό το ότι στο έτος της Ιθαγένειας ε, υπάρχουν τέτοιες περικοπές ε, που είναι σχεδόν απίστευτο. Αυτό πια είναι και παράλογο. Γι' αυτό λοιπόν την επιστολή που συζητήσαμε χθε ε, στις συνεδρίες των συντονιστών θα τη συντάξω και νομίζω ότι όπως και εσείς μας το προτείνατε θα είμαστε αυστηροί διότι νομίζω ότι χρειαζόσαστε ένα έγγραφο για να μπορείτε να εργαστείτε. Δεν πρόκειται για την θέληση αυτής της Επιτροπής, αλλά πρόκειται για το ότι είναι ορισμένα πράγματα απαραίτητα για την επόμενη γενιά. Εδώ και 7 χρόνια δουλεύουμε σε θέματα εκπαίδευσης, παιδείας, κατάρτισης, ε, πολύ σημαντικά θέματα. Αυτή είναι η ψυχή της Ευρώπης και σε αυτή την ψυχή διαγράφουμε τα κονδύλια. Δεν είναι δυνατόν. Ε, η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει να αγωνιστεί μαζί μας γιατί η Κομισιόν στη τελική ανάλυση και αυτή δεν είναι ιδιαίτερα γενναιόδρη. Με το 75% αύξηση ε, των ε, κονδυλίων δεν ξεπέρασε κάποια, κάποιο όριο αλλά προσπάθησε να κάνει κάτι το οποίο είναι σχετικά σωστό. Και νομίζω λοιπόν ότι αν φτάναμε στο 75% θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Αλλά ξέρετε πόσο δύσκολα είναι όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισηγησή σας. Ε, θα επανέλθουμε. Οι διαπραγματεύσει θα ξεκινήσουν το Μάιο. Ε, και εδώ είμαστε λιγάκι μεταξύ σκύλας και χάριδος. Ε, ε, μιλάμε για πράγματα που δεν θα πρέπει να μιλάμε γιατί δεν έχουμε λεφτά. Αυτό δεν μου έχει συμβεί ποτέ σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι ευρωβουλευτής. Ποτέ δεν ήταν τα πράγματα όπως είναι σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτομαι πραγματικά πού καταντήσαμε. Και αν σκεφτώ ότι ε, εφέτος ε, το θέμα ε, των πληρωμών και των υποχρώσεων αποκλίνει τόσο πολύ, τότε ξέρω τι θα γίνει. Βεβαίω και θα πληρώσουμε, αλλά θα πληρώσουμε με χρήματα που είναι για το μεθεπόμενο χρόνο εγώ δεν μπορώ να έχω τέτοιο δυσπροπολογισμό προπολογισμό. Πώς, θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να επανέλθει η τάξη και στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν για να μπορούμε να ε, παρουσιαστούμε και απέναντι στους ε, ψηφοφόρους μας, οι οποίοι βέβαια ποτέ δεν τα έχουν καταλάβει γιατί και ποτέ δεν τους το είπανε. Ποτέ δεν τους είπαν ότι αυτό που έχουμε κατ' ουσίαν δεν είναι νομοθετικό έγγραφο. Είναι ένα έγγραφο ε, το οποίο το σκέφτηκαν κάποιοι, αλλά κατ' ουσίαν είναι μόνο έγγραφο εργασίας και τίποτα άλλο. Όταν όμως έχουμε εκλεγεί πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και όχι αυτό που λένε πολλοί ότι το κοινοβούλιο θέλει όλο συνεχώς λεφτά. Εμείς θέλουμε τα λεφτά που έχουμε να τα δαπανάμε σωστά. Ο κύριος Λόκαγκάρτ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ήδη είπατε ότι είναι δύσκολο να το συζητήσουμε αυτό σε τόσο πρώιμο στάδιο. Θα προσπαθήσω να το κάνω παρόλα αυτά με κάποιες παρατηρήσεις. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα ε, προγράμματα της Επιτροπής μας είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε την Creative Europe, έχουμε την Ευρώπη για τους πολίτες, έχουμε τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης και βεβαίως ε, θα χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να πω ότι για να επιτύχουν τα προγράμματα αυτά πρέπει να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Θέλω να το τονίσω αυτό γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο φαντάζομαι ότι δεν μιλάμε και για πολλά λεφτά. Οπότε είμαστε πιο ευάλωτοι βέβαια στην Επιτροπή μας με τα προγράμματά μας και ε, αν δούμε για παράδειγμα τι περικοπές ε, υπάρχουν, εμείς είμαστε μάλλον αυτοί που υποφέρουμε περισσότερο και θα ήθελα να δω κάποια από τα αριθμητικά στοιχεία που θα μας παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, πάντως σύμφωνα με αυτά που έχω δει 20-25% σε κάποιες γραμμές προπολογισμού. Είναι άσχημα τα πράγματα δηλαδή για μας και θέτει το ζήτημα του κατά πόσο τα νούμερα αυτά πρέπει να τύχουν διαπραγμάτευση όντω ή αν ε, βρισκόμαστε σε μια παγιωμένη, ενώπιον μιας παγιωμένης κατάστασης. Ε, είπατε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι συνομοθέτης, δεν είναι νομοθέτης και αυτό φαντάζομαι ότι αφήνει κάποιο περιθώριο ε, ελιγμών, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο περιθώριο έχουμε για τη διαπραγμάτευση των, διαπρα... των, ε, των γραμμών αυτών προϋπολογισμού, γιατί έχω λιγάκι μπερδευτεί την τελευταία, μετά την τελευταία συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχαμε την εντύπωση ότι οι γραμμές προπολογισμού είχαν οριστεί και ότι εμείς ε, πρέπει να αποδεχθούμε απλώς ε, τις συνέπειες. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό και θα ήθελα να μου πείτε και τη δική σας άποψη. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι στον τομέα του αθλητισμού είναι ένα νέο πρόγραμμα και βεβαίως πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για τον αθλητισμό, και βεβαίως πρέπει να το κάνουμε αυτό και νομίζω ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην ε, ε, το παραγνωρίσουμε, να υπάρξει επαρκή χρηματοδότηση και γι' αυτό όσον αφορά τώρα τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε και η Πρόεδρος, να αρχίσει η δουλειά τώρα για να μπορέσουμε να υποβάλουμε κάποια προγράμματα μέχρι τα τέλη Μαΐου για τις ε, τρέχουσες προπαρακευαστικές δράσεις και προγράμματα που θα ισχύουν και το 2014 πρέπει να τα επανυποβάλουμε. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες από τώρα, αλλά βέβαια θα κάνω ένα σχέδιο για, το... για τα νέα ε, προγράμματα που τα δρομολογούμε σήμερα, σήμερα ξεκινάνε, που φαίνονται να ξεκινούν καλά και θα θέλαμε η πλειοψηφία νομίζω της Επιτροπής μας να συνεχίσει και το 2014. Το ερώτημά μου προς εσάς κυρία ε, Γένσεν αυτό είναι και θα ήθελα να με διαφωτίσετε όσο μπορείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα. Η Άννα Γένσεν και εγώ συνεργαζόμαστε στην Επιτροπή προπολογισμού και είμαστε πολύ εξοικειωμένε με όλες τις εξελίξεις. Συμφωνώ λοιπόν με την Τόρες ότι η κατάσταση πραγματικά είναι χειρότερη από τα προηγούμενα χρόνια. Και είπε και η Άννα ότι οι πληρωμές ε, έχουν πλέον είναι ε, θέμα πολιτικής επαφής. Τα προηγούμενα χρόνια εμείς ασχολούμεθα με το επίπεδο των πιστώσεων, υποχρεώσεων, διότι ξέραμε ότι μετά θα γίνουν πραγματικότητα με τις πληρωμές. Τώρα σταμάτησε αυτή η προσέγγιση. Αν δεν καλείς τι έγινε την έκτακτη σύνοδο κορυφής το Φεβρουάριο και τι αποφάσεις πήρε το Συμβούλιο, υπάρχει μία καταστροφική διαφορά 20 δις μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών. Θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπες για την πολιτική κοινωνία μεταξύ μας. Και εμείς ως Επιτροπή και εσείς ως πρόεδρος εκ μέρους της Επιτροπής μας ίσως θα πρέπει να κάνετε δημοσίως μια ανεξή λέγοντας ότι είμαστε απόλυτα δυσαρεστημένοι με τον προϋπολογισμό που έχουμε μπροστά μας. Ίσως ο αντίκτυπος δεν θα είναι πολύ σημαντικός αλλά ας το κάνουμε τουλάχιστον. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε τους πολίτες να καταλάβουν ότι δεν είναι θέμα συμφερόντων του καθενός, αλλά συλλογικά κάτι μας ενδιαφέρει. Και έτσι θα έχουμε το πράγμα το 2020. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι πολλές χώρες μας έχουν προβλήματα στον κρατικό προϋπολογισμό τους. Είναι μεγάλο όμως το πρόβλημα το ότι κάνει πιο πολλές περικοπές στον κοινοτικό προπολογισμό παρά στου εθνικού στο Συμβούλιο. Σε όλη αυτή την ε, ανακίνηση που γίνεται με την πολιτική χρειά ότι κόβουμε τον ε, κοινοτικό προπολογισμό για να μην κάνει περικοπές στου εθνικού, είναι μπλα μπλα. Και όπως βλέπετε, όλο και περισσότερες ανισορροπίες δημιουργούνται και όλο και περισσότερο, συγγνώμη, όλο και λιγότερο όλοι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να γίνει σε κοινοτικό επίπεδο. Τώρα, υπάρχουν και άλλα θέματα με πολιτική σημασία και χρειά. Ξέρετε ότι το Συμβούλιο κάπου έχει κάνει κάποιες μικρές αυξήσεις, όπως λέει, στην παιδεία και στην κουλτούρα. Αλλά αυτό είναι ένα τρίκ και πάλι, διότι και η Κομισιόν και η Επιτροπή ήθελαν να δώσουν στο πρώτο κεφάλαιο και στην παιδεία κάποια συμπληρωματικά κονδύλια, αλλά κάνουν συγκρίσεις των αριθμών που περικόπτουν. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει είναι να συγκρίνουμε τι είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή και, και πού καταλήξαμε στο τέλος. Εδώ έχετε λοιπόν τρομερές περικοπές και θα πρέπει να το δούμε πολιτικά αυτό το θέμα. Το ίδιο έγινε και με το Europe for Citizen. Πολύ κακέ εξελίξει σε ένα τομέα στον οποίο πάντα λέγαμε και έλεγε και το Συμβούλιο πρέπει να προσεγγίσουμε τους πολίτες, πρέπει να τους δώσουμε δυνατότητες να έρθουν σε επαφή με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά την άποψή μου είναι ποντί κοντόφθαλμη και συντηρητική αυτή η προσέγγιση του Συμβουλίου όσον αφορά ε, τις ε, ε, μελλοντικές, τις τωρινές και μελλοντικές χρηματοδίτες. Θα πρέπει λοιπόν να στείλουμε μία επιστολή στον Λαμασούρ λέγοντας ότι το μπορούμε να τον εξοδοτήσουμε, να κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους εκτός των τυχών, γιατί είναι κρίμα να γίνονται αυτά που γίνονται. Ευχαριστώ η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω κάποια πράγματα. Να σας δώσω κάποιες ε, πληροφορίες. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εμείς ασχολούμαστε με διάφορα θέματα, με τη νεολαία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, αλλά στηρίζω αυτά που είπε η Ντόρις ε, για το πρόγραμμα Εράσμους. Για μας ε, αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι έχουμε ε, προβλήματα χρηματοδότησης και θα χαιρόμαστε να μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, ότι κάθε χρόνο να εξηγούμε ότι υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότηση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι το πιο επιτυχημένο ε, πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για 25 εκατομμύρια νέους ε, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό και κατόπιν τούτου ε, θα πρέπει να είναι αντάξια η ενασχόλησή μας. Είναι το πιο επιτυχημένο μας πρόγραμμα έχει προσφέρει μεγάλη υπεραξία. Το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 προβάλλει το ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτά τα προγράμματα να στηρίζονται. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάει κανείς για αριθμούς ε, που δεν υπάρχουν. Όλα αυτά είναι λιγάκι αφηρημένα αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να αγωνιστούμε ε, κατά ε, της εγκατάλειψης του σχολείου. Μόνο εφόσον υπάρχει εκπαίδευση μπορούμε να ε, στηρίξουμε τα πανεπιστήμια. Χρειαζόμαστε χρήματα για πανεπιστημιακά προγράμματα για να μην εγκαταλείπουν τα παιδιά το σχολείο. Τώρα, πώς βλέπετε εσείς την υποστήριξη των νέων. Υπάρχει μια νέα πρωτοβουλία εκ μέρους της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, γνωρίζω ότι όλα αυτά σχετίζονται με ε, και μέτρα για την απασχόληση. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σας επί του θέματος. Το λόγο έχει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Um, Θα ήθελα να κάνω κάποιες διευθυντικές παρατηρήσεις όσον αφορά τη θέση της Κομισιό. Πρώτα απ' όλα, τέλος Μαρτίου η Επιτροπή ενέκρινε μια τεχνική προσαρμογή, όπως ονομάζεται. Δηλαδή, κάποιες αλλαγές στις προτάσεις που κάναμε για το πολιετές, βάσει των ε, αριθμό ο οποίος συμφώνησε το Συμβούλιο τον Φεβρουάριο. Και υπενθυμίζω για το κεφάλαιο 1α. Περικοπή 50% σε σχέση με την αρχική πρόταση. Και αυτό είναι το ποσοστό που προτείνεται να περικοπεί. Κεφάλαιο 3. Γενικά. 16,6% Creative Europe 19%. Διότι εδώ υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί στους οποίους θα είναι πιο περιορισμένες ε, οι περικοπές για τεχνικούς λόγους. Ίσως κάποια λόγια για την ε, ετήσια κατανομή. Άκουσα με μεγάλη σαφήνεια αυτά το επίπεδο για το σφαιρικό πολιτικό πλαίσιο στο οποίο κινηθήκαμε. Στην Επιτροπή όμως πρέπει να σκεφτούμε την ετήσια κατανομή των ποσών. Και μία γραμμική εφαρμογή των μειώσεων για την Creative Europe θα μας είχε οδηγήσει σε μείωση του προϋπολογισμού για το 14-15-16 σχέση με το 2013. Στην πρόταση της Επιτροπής του, του Μαΐου αντιμετωπίζεται το πρόβλημα αυτό εν μέρη, άρα έχουμε μειωμένη ε, μείωση το 14, σχεδόν καμία μείωση το 15, αλλά θα ήθελα το πρόβλημα αυτό να το αναφέρω ιδιαίτερος και να το επισημάνω. Είναι θέμα εφαρμογής για το μέλλον του προγράμματος Creative Europe και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περαιτέρω συνολικά. Ενώ προφανώς στην Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Κουλτούρα να συμμεριζόμαστε τις παρατηρήσεις θα ήθελα να τονίσω ότι μετά από τις περικοπές που πρότεινε στις τεχνικές προσαρμογές η Επιτροπή, ακόμη εξετάζουμε τα πράγματα σε σταθερές τιμές για την αύξηση χρηματοδότησης της παιδείας και της κατάρτισης των νέων με αύξηση 47% σε σχέση με την, τους τρέχοντες ε, ρυθμούς, οπτικοακουστικά μέτρα 9% και τελικά δύο λόγια για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Προσπαθήσαμε να τα ενσωματώσουμε στο μέτρο του δυνατού στη νομική βάση του Εράσμους για όλους και Creative Europe και ίσως αυτά είναι τα δύο καλύτερα παραδείγματα τα οποία έχω να σας πω για τα θέματα και αθλητισμού και όλους λοιπόν. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Κρέσε, δεν σας ε, καταλαβαίνω πραγματικά, μάλλον επειδή και εσείς ε, δεν νιώθετε καλά στο πεσί σας με αυτά που λέτε. Ε, ειλικρινά δεν μπόρεσα να σας παρακολουθήσω. Ίσως να φταίω εγώ, αλλά και η παρακαθήμενη μου ούτε και τι κατάλαβε αυτά που λέτε. Ε, ίσως να πρέπει να τα πλουστεύσουμε λιγάκι για να καταλάβουν όλοι περί τίνος πρόκειται. Αν δει κανείς τα στοιχεία που μας στείλετε, τι προκύπτει. Ανάμεσα σε αυτά που προτείνει η Επιτροπή, δηλαδή 72% αύξηση, τώρα με βάση αυτά που πρότεινε το Συμβουλίο, προτείνετε εσεί αύξηση μόνο 47%. Καλά, το κατάλαβα αυτό. Αυτό καλά. Πάμε τώρα στην Creative Europe. Και εκεί τα μπερδέψαμε. Μπερδευτήκαμε τελείω. Είπατε 34% είχατε προτείνει και τώρα φτάσαμε στο 19%. Μα τι είναι αυτά. Και τι να κάνουμε τώρα με την Creative Europe. Είχαμε πει 34% και φτάσαμε στο 9% δεν ξέρω, αυτό δεν γίνεται. Εσείς κάνετε μόνο υπολογισμούς, εσείς δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να βγάζετε σε αριθμούς αυτά που σας λέει το Συμβούλιο. Και μετά ερχόμαστε στην Europe for Citizens. Ξέρω ότι δεν είστε αρμόδιος για αυτό, αλλά εκεί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Εκεί έχουμε ακόμα και μείον 23%, όπως εσείς είχατε προβλέψει μείον 5%. Τι να σας πω, ε, κανείς δεν μπορεί να τα δεχτεί αυτά τι νόημα έχει τώρα να συζητάμε. Εσείς δεν μπορείτε να τα αλλάξετε. Ο μόνος που μπορεί να τα αλλάξει είμαστε εμείς, Γιάννησεν Τρούπελ, Επιτροπή Προπολογισμών. Πρέπει να δώσουν μάχη για να αλλάξουν οι αριθμοί, γιατί αλλιώς ε, γινόμαστε φεδροί. Ε, Βεβαίω ε, θα κάνω μια συνέντευξη τύπου, όχι ότι θα γίνει τίποτα και ότι θα βάλω κόσμο στα κλάματα. Βέβαια το Twitter βοηθάει λίγο, το Twitter έχει κάποια αποτελεσματικότητα. Από την 1η Ιουλίου θα έχουμε άλλη μια χώρα που θα προσχωρήσει και αυτούς πρέπει να τους ταΐσουμε κάπως. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν. Πώς οι κύριοι και οι κυρίες, και οι κυρίες φοβάμαι αυτά είναι οι κυρίες, πώς τα παρουσίασαν όλα αυτά. Λοιπόν, εμείς δεν τα εγκρίνουμε, θα αγωνιστούμε, Λαμασούρ Γένσεν, ε, θα τους ε, παρακινήσουμε που δεν χρειάζεται και πολύ προσπάθεια και αυτοί τα ίδια σκέφτονται. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω να πείτε στην Κομισιόν ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, που μας ε, είπαν ε, ποια είναι η άποψή του, αλλά μπορούν και αυτοί να θεωρούν ότι εμείς δεν θα τα δεχτούμε. Νομίζω ότι εδώ να κλείσουμε τη συζήτηση. Αν θέλετε να δώσω το λόγο στην κυρία Γένσεν, αλλά τώρα τι θα συζητάμε. Α, κι άλλος. Ποιος άλλος θέλει το λόγο. Η κυρία Ίναϊσεν είναι εδώ. Η κύριος, κύριος, κυρία. Αλλά νομίζω ότι τα έχω πει ε, λέγοντας ε, πόσο κακή είναι η Citizens for Europe. Εκπροσωπώ την κυρία Ινάιχεν, Δεν έχω να σας πω τίποτε πέρα, πέρα από αυτά που ξέρετε. Δεν μπορώ να σας δώσω την πρότασή μας, γιατί το σχέδιο προϋπολογισμού δεν έχει ακόμη υποβληθεί. Δεν έχει περάσει από το Σώμα των Επιτρόπων. Όλα όσα μπορούμε να σας ε, πούμε, τα γνωρίζετε ήδη. Θα δείτε για τους Europe for Citizens, για τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας. Ε, ναι, έχει υπάρξει σοβαρή μείωση εκεί. Και δεν ε, είναι πολύ καλά τα πράγματα. Δεν μπορώ όμως να σας πω τίποτε παραπέρα. Δεν μπορώ να σας δώσω όλα τα νούμερα για όλες τις γραμμές προϋπολογισμού. Αλλά θα έχετε την πρότασή μας στη διάθεσή σας ε, σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τώρα θα, κάνω, θα, γίνω κακιά, αλλά να σας πω το εξή. Θα ευχόμουν η κυρία Ρέντινγκ να αγωνιστεί ε, με το ίδιο πάθος ε, για τη δική μας υπόθεση όπως αγωνίζεται για τις ποσοστώσεις των γυναικών. Εκεί κάτι μπορεί να κάνει. Ε, βέβαια σε άλλες περιπτώσεις εξαρτάται και από άλλους. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι από κοινού. Ούτε η κυρία Ρέντινγκ παραπονέθηκε για αυτές τις περικοπές του 23%. Να της πείτε χαιρετίσματα, αλλά θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν και εκείνη όπως και εγώ έβγαινε να κάνει συνέντευξη τύπου. Εμείς τη στηρίζουμε όταν εκείνη διαμαρτύρεται. Να μας στηρίξει και αυτή τώρα. Και ευχαριστώ κύριε Μπέκερ που με χειροκροτάτε. Εντάξει, δεν ήταν απαραίτητο, αλλά χάρηκα παρόλα αυτά. Κυρία Γιάννη, έχει το λόγο. Yes, thank Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και εγώ είμαι στη διαπραγματευτική ομάδα για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για αυτό το λόγο. Ε, τέθη το ερώτημα κατά πόσο τα νούμερα των αριθμών κρατών, των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων είναι αυτά τα οποία επεξεργαζόμαστε. Μπορούμε να δούμε βέβαια από τις συζητήσεις και από τις διαπραγματεύσεις ε, την τελευταία φορά που είχαμε πολιετές ε, δημοσιονομικό ε, πλαίσιο, είχαμε 5 δισεκατομμύρια για 7 χρόνια. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε υπεραισιόδοξοι σε σχέση με το πόσο ποσό που θα μπορούσαμε να έχουμε ε, επιπλέον από αυτό το ποσό, όμως τα ποσά τα οποία ζητάτε στην ε, Επιτροπή σας, ε, στην ευρύτερη, στο ευρύτερο πλαίσιο δεν είναι τεράστια και ειδικότερα όταν βλέπουμε ότι υπάρχει καλή εφαρμογή, όταν αξιοποιούνται πράγματι τα κονδύλια, είναι τόσο το καλύτερο. Μπορείτε να αποδείξετε ότι είναι καλά τα αποτελέσματα των προγραμμάτων. Νομίζω λοιπόν ότι πραγματικά είναι δίκαιος ο αγώνας σας και μπορείτε να τον προωθήσετε. Βέβαια, οι βασικές περικοπές που είδατε σε νούμερα, σε πραγματικούς αριθμούς, είναι στις πολιτικές ε, γεωργίας και συνοχής. Εκεί υπήρξαν τεράστιες ε, περικοπές για τις, ε, στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν υπάρχει κανένα απολύτως, δεν υπάρχει καμία διαμάχη ως προς αυτό γιατί υπήρξαν οι, οι περικοπές αυτές, οπότε παρακαλώ να συνεχίσετε τον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω. Για μας ο προϋπολογισμός ήταν πάντα μικρός διότι εμείς είμαστε αρμόδιοι για πολλά θέματα επικουρικά. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν το μικρό το κάνω ελάχιστο, καταλαβαίνετε ότι πια δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το μικρό ποσό, το οποίο θα μας ε, αφαιρέσετε, για μας είναι μεγάλο. Αυτό λοιπόν αν ε, το αφαιρούσα κανείς από τα διαρθρωτικά ταμεία, ούτε καν θα το πρόσεχαν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βλέποντας λοιπόν τώρα ότι έχουμε προβλήματα με το πρόγραμμα Erasmus, ξέρετε γιατί τα έχουμε τα προβλήματα, διότι ε, για πολλά έτη ε, από τα διαρθρωτικά ταμεία και από τα γεωργικά ταμεία δεν υπήρξε ανάκληση κονδυλίων και οι, ε, τα κράτη-μέλη κράτησαν αυτά τα κονδύλια. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο δοχείο όπου μπαίνουν κονδύλια και από την άλλη να τα παίρνουμε. Κάθε χρόνο θα πρέπει να βλέπουμε ε, τι μας αντιστοιχεί και εμείς δεν μπορούμε να ε, δαπανίσουμε διαρθρωτικά κονδύλια. Γι' αυτό λοιπόν τα χρήματα τα οποία δικαιούμαστε χάνονται αυτό όμως ε, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε στον ε, απλό πολίτη. Ξέρετε, στο ε, Στρασπούργο, επειδή εκεί από την περιοχή είμαι εγώ, έρχονται πολλοί επισκέπτες και πραγματικά πολλοί τα έχουν ψηλιαστεί όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι που κάναμε σήμερα τη συζήτηση και θα παρακαλέσουμε και την κυρία Ρέντινγκ να μας στηρίξει και αυτή ανοιχτά. Και νομίζω ότι και οι κύριοι και οι κυρίες ε, της ε, ε, διεύθυνση εκπαίδευση και ενόλα και αυτή μας την και η κυρία Βασιλείου να ανοίξει και αυτή το στόμα της δεν νομίζω ότι έχει νόημα αυτή να τα δέχεται όλα νομίζω ότι πρέπει να αγωνιστούμε και χρειαζόμαστε κοινό μέτωπο σε αυτό τον αγώνα ευχαριστούμε τους Γένσεν, Τρούπελ και Λόκεγκαρ πάει αυτό το 11 της μερίσιας διάταξης την εσωτερική αγορά την κλείσαμε. Πάμε στο επόμενο θέμα, στην αναθεώρηση της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ. Ανασχεδιασμός. My language, so if you can use your headsets, please. Thanks. Vážení kolegovia, ďakujem veľmi pekne, že som dostala príležitosť byť spravodajcom tejto veľmi dôležitej správy o reforme vzdelávania. Sa ευχαριστώ pára poli, που είμαι εισηγήτρια για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Καταρχήν θέλω να πω ότι η έκθεση Επιτροπή είναι πολύ καλή, αποτελεί μια πολύ καλή βάση ε, που θα μας ε, χρησιμεύσει. Γιατί λοιπόν πρέπει να ασχοληθούμε με την πολιτιστική ε, μεταρρυθμίση. Έχουμε τεράστια προβλήματα με την ανεργία των νέων. Αν θέλετε η γαλλική καμπίνα... Ναι, Λοιπόν, εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ με τρία θέματα. Το μέλλον της ε, νεολαίας, τις συνεργασίες και την εκπαίδευση των ενηλίκων. Η ανεργία των νέων είναι 23,5%. Αυτά είναι τα στοιχεία του Μαρτίου. Ε, παράλληλα όμως ε, έχουμε και 2 ε, εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό λόγω του ότι δεν έχουμε αρκετούς εκπαιδευμένους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Οι δεν συμμετέχουν τόσο στην επαγγελματική κατάρτιση και εάν δεν θέλουμε να έχουμε μία χαμένη γενιά, πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Εγώ λοιπόν συμφωνώ ότι η ανεργία των νέων μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της εκπαίδευσης. Βέβαια η διαδικασία αυτή είναι ε, μακροχρόνια, δεν μπορεί να γίνει μια νυχτή. Και βεβαίως δεν πρόκειται μόνο για τις ε, επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, ε, πρόκειται και για την, για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι νέοι πρέπει να έχουν τις δυνατότητες για να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Τι είναι όμως πιο σημαντικό πιο σημαντικό είναι οι δεξιότητες για την αγορά εργασίας ή είναι σημαντικό οι νέοι να μπορούν να βρουν το επάγγελμα που ονειρεύονται. Σήμερα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να εξασκήσει κανείς το επάγγελμα που είχε ονειρευτεί. Γι' αυτό λοιπόν τώρα πλέον ε, πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με το να ενταχθούν οι νέοι στην αγορά εργασίας. Έχω και άλλα θέματα που επιθυμώ να επεξεργαστούμε. Η ε, Κομισιόν, παραδείγματος χάρη, ε, προτείνει κάποιες ε, δεξιότητες για τους νέους. Παραδείγματος χάρη, προαγωγή της κινητικότητας των νέων. Νομίζω ε, είναι σωστό αυτό να ληφθεί υπόψη κατόπιν εκμάθηση ξένων γλωσσών. Υπάρχουν κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι ξένες γλώσσες ε, είναι σχεδόν ε, ανύπαρκτες. Οι Γαλλία, ας πούμε, δεν μαθαίνουν πολλές ξένες γλώσσες οι Γάλλοι, αλλά υπάρχουν και άλλα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Επιπλέον, στο εγγύς μέλλον δεν θα έχουμε και μεταφραστές με αγγλικά μητρική γλώσσα, γιατί ε, οι Εγγλέζοι δεν μαθαίνουν καμία ξένη γλώσσα. Επίσης ε, πρέπει να δούμε τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι νέοι χρειάζονται επιχειρηματικές ε, ικανότητες όταν δεν είναι σε θέση να βρουν θέση εργασίας πρέπει να είναι σε θέση να ιδρύσουν ε, μόνοι τους μια επιχείρηση και να προσφέρουν απασχόληση και σε άλλους. Αυτή είναι μια ε, προληπτική προσέγγιση κατόπιν όσον αφορά την προαγωγή του πολιτισμού και όλα τα άλλα προφανώς και τα στηρίζουμε όλα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η προαγωγή της επαγγελματικής ε, εκπαίδευσης. κρατημέλη έχουν το σύστημα της ε, ε, γενικής κατάρτισης τα γυμνάσια, πούμε, και τα λύκεια, αλλά αν έχει κανείς ε, απολυτήριο λυκείου, δεν έχει συγκεκριμένες ε, δεξιότητες, πρέπει να πάει στο πανεπιστήμιο να φοιτήσει ή ε, σε κάποια ειδική επαγγελματική σχολή. Γι' αυτό, λοιπόν, χρειαζόμαστε τέτοιου είδους ειδικέ επαγγελματικές σχολές. Έχω δει διάφορα στατιστικά δεδομένα και είναι σαφές ότι πολύ σύντομα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειάζεται 900.000 ε, νέους ε, με γνώσεις πληροφορικής. Εάν λοιπόν σε πέντε χρόνια θέλουμε να έχουμε τόσους πολλούς ανθρώπους με γνώση πληροφορικής, πρέπει ήδη να αρχίσουμε τώρα. Πρέπει ήδη τώρα οι άνθρωποι αυτοί να αρχίσουν να σπουδάζουν πληροφορική. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να προάγουμε την επαγγελματική κατάρτιση. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά, γιατί η πληροφορική είναι ένα τομέα που εξελίσσεται ταχύτατα. Ως προς την επαγγελματική κατάρτιση υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις. Στη δική μου τη χώρα η τεχνική κατάρτιση ε, θεωρείται υποδέστερη της ε, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί αν χρειαστεί κάποιο σπίτι του να επισκευάσει κάτι, χρειάζεται έναν ειδικό. Χρειαζόμαστε λοιπόν τους τεχνίτες και όχι μόνο αυτούς με ευρύες επαγγελματικέ ή μάλλον ε, εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Καλό θα ήτανε να υπάρχουν σύμβουλοι επαγγελματικής κατάρτισης έτσι ώστε να μην πιστεύουν οι γονείς ότι το παιδί τους πρέπει να σπουδάσει μόνο γιατρός ή δικηγόρος. Υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ιστοσελίδα που είναι πάρα πολύ καλή σχετικά με τις δεξιότητες, μπορείτε να την επισκεφτείτε και εκεί υπάρχουν πολλές και χρήσιμες πληροφορίες. Στο μέλλον θα επικρατήσει εξή τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα χρειαζόμαστε όλο και περισσότερους ε, εκπαιδευμένους, εργαζόμενους. Βεβαίως και θα παραμείνει ε, παραμείνουν τα χειροτεχνικά επαγγέλματα. Ο συνάδελφος Φίσερ ε, πάντα λέει ότι χρειαζόμαστε και τους παραδοσιακούς τεχνίτες. Και αυτό κατά την άποψή μου είναι μια πολύ καλή ιδέα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι το εξής. Ένας ε, κάθε τρίτος μάλλον Ευρωπαίος εργοδότης ή εργαζόμενος μάλλον είναι ή έχει περισσότερα ή λιγότερα επαγγελματικά προσόντα. Άρα πολλοί εργαζόμενοι ε, δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χρειαζόμαστε διάφορα επαγγέλματα. Πολλές φορές ε, γίνεται λόγος για αγύρανση της Ευρώπης και γι' αυτό χρειαζόμαστε και απασχολούμενους ε, ε, σε αυτό το τομέα της ε, υγείας. Βεβαίω ανάλογες πρέπει να είναι και οι απολαβές που προσφέρονται. Άλλο σημαντικό θέμα. Η συνεργασία με τα μορφωτικά ιδρύματα και συσχετισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και αγοράς εργασίας. Και αυτό πρέπει να το στηρίξουμε. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά στη Γερμανία και την Αυστρία. Πρέπει λοιπόν να προσφέρουμε τη δυνατότητα στους φοιτητές ε, να συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής εξάσκησης και μετά το τέλος ε, του σχολείου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας εδώ λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, προβλέπει τη δυνατότητα αμοιβόμενων ε, μαθημάτων πρακτικής εξάσκησης. Όσον αφορά τώρα την αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, πολλά χρόνια γίνεται αυτή η κουβέντα, δεν ε, έχει προχωρήσει βέβαια και θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται δυστυχώς στο μηδέν. Και αυτό περιορίζει την κινητικότητα των εργαζομένων. Θα ήταν ευπρόσδεκτο λοιπόν αν ε, λειτουργούσε η αναγνώριση των δεξιοτήτων. Και όσον αφορά την εκπαίδευση ε, των ενηλίκων, χαίρομαι που ε, προβάλλεται η διαβίου Πράγματι, οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε θέση να αποκτούν νέες δεξιότητες και μόνο με τον τρόπο αυτό θα προσαρμοστούν στις ε, μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς-εργασίας. Να πω κάτι για την επαγγελματική κατάρτιση των δασκάλων. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί πολύ σημαντική, ιδιαίτερα σημαντική προϋπόθεση. και οι δάσκαλοι πρέπει να ε, εκπαιδεύονται. Εάν δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι οι καθηγητές και οι φοιτητές δεν μπορούν να σημειώσουν πρόοδο. Και όσον αφορά τις ε, συνεργασίες, ανέφερα ήδη ότι πρόκειται για τη συνεργασία ανάμεσα ε, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και την αγορά εργασίας. Πρέπει να υπάρχει προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Βεβαίως ε, τα πανεπιστήμια εδώ και αιώνες είναι ανεξάρτητα και δεν το αμφισβητώ, όμως τα πανεπιστήμια θα πρέπει να σκεφτούν κατά πόσον αυτά που διδάσκουν είναι προσαρμοσμένα στην πραγματικότητα. Η φίτηση δεν είναι αυτός σκοπός πρέπει να έχει κανείς δυνατότητα να επιβληθεί στην αγορά εργασίας. Επίσης η άτυπη εργασία νομίζω είναι πολύ χρήσιμη για τους νέους οι οποίοι αποκτούν ε, πολύ χρήσιμες εμπειρίες. Είναι και αυτό μια σημαντική συνεισφορά για τους νέους όπου οι νέοι συναντώνται και με ανθρώπους από άλλους ε, πολιτισμούς. Ε. Η άτυπη εκμάθηση είναι λοιπόν πολύ σημαντική. Έχω πάρα πολλά ε, να σας πω, δεν μπορώ να σας τα πω όλα, αλλά Βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις ε, ερωτήσεις σας. Ε, τέλη Μαρτίου οργανώσαμε μια στρογγυλή τράπεζα. Εκεί συμμετείχαν 23 διαφορετικοί φορείς. Ευχαριστώ πολύ για την οργάνωση και αυτά που είπα τώρα κατ' ουσίαν είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων της ε, στρογγυλής τράπεζας όπου εκπροσωπήθηκε και ο ιδιωτικός τομέας και άλλοι φορείς της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 7 Μαΐου θα λάβει χώρα η επόμενη στρογγυλή τράπεζα και προσβλέπω στη συμμετοχή σας. Ελπίζω να μην μίλησα πολύ γρήγορα. Nein, wir haben es gut äh, äh, Όχι, όλα εντάξει. Κατερίνα, αν σκεφτεί κανείς την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης, θυμάσαι, είχαμε πει και τότε, ξέρουμε ότι χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα αλλά δεν θα ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επέλεξαν αυτό το φρικτό προϋπολογισμό ε, δεν ε, τα είχαν σκεφτεί όλα αυτά νωρίτερα. Ε, ελπίζω να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε. Ελπίζω ότι η διαδικασία αυτή τη φορά θα πάει καλύτερα και θέλουμε η διαδικασία της Μπολόνιας να πάει καλύτερα, να προωθήσει την κινητικότητα, κάτι που δεν συμβαίνει για την ώρα. Σε τρία χρόνια πρέπει να μάθει κανείς αυτά τα οποία κανονικά θα μάθαινε σε πέντε. Η διαβίου εκμάθηση είναι για τους φοιτητές και όχι για τους διδάσκοντες. Καταλαβαίνω τι εννοείτε. Έχετε το λόγο. Η άποψή μου είναι ότι η επένδυση σε δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα ε, έρχεται τουλάχιστον με 10 χρόνια καθυστέρηση. Έχουμε ασχοληθεί με άλλα πράγματα, προκλήσεις, προτεραιότητες, ε, ε, στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η οικονομική κρίση ε, μας υποχρέωσε να το εγγράψουμε στην ημερήσια διάταξη και όντως έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η εκπαίδευση δεν είναι εξαιρετική σημασίας, ε, ε, για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ε, της ε, οικονομίας ε, της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο. Να τονίσω κάτι μόνο. Πρέπει να μειώσουμε, και συμφωνώ με ε, τους υπόλοιπους συναδέλφους, πρέπει να μειώσουμε το κενό ανάμεσα στην, ε, στις επιχειρήσεις, στην επιχειρηματικότητα και στην εκπαίδευση. Πώς να το κάνουμε αυτό περισσότερα δημόσια κονδύλια δεν θα μπορούσαν ε, να αποτελέσουν την ε, σωστή απάντηση. Επίσης, η συζήτηση για τη δημόσια χρηματοδότηση ε, στην εκπαίδευση είναι δύσκολη. Δεν υπάρχουν πλέον τέτοιου είδους δημόσια κονδύλια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι, καταρχάς, η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας χρηματοδότησης για την εκπαίδευση και επίσης εξέβρεση νέων προσεγγίσεων, νέων νέων τρόπων αύξησης της αποτελεσματικότητας ε, των δαπανών ε, για την εκπαίδευση. Να αναλύσουμε την ε, πιθανότητα αύξησης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην εκπαίδευση εγώ ως όδης εισηγητής ε, με χαρά θα συνεργαστώ με την εισηγήτρια, την κυρία Νεβεντάλοβα, όπως επίσης και με τους υπολείπους συναδέλφους στην Επιτροπή μας, για ένα πολύ σημαντικό θέμα, μια πολύ σημαντική έκθεση για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Εισηγητρία, σήμερα μας παρουσιάσατε την δική σας ε, άποψη για το πρόβλημα αυτό. Επί της ουσίας συμφωνώ απολύτως με την έκθεσή σας, διότι πιστεύω ότι όλα αυτά τα οποία λέτε είναι πολύ θετικά, πολύ γόνιμα. Θα πρέπει επίσης να συγχαρούμε για αυτή την ε, πρωτοβουλία την Επιτροπή. Έπρεπε να γίνουν τα πράγματα όπως είπε και η Επιτροπή νωρίτερα, αλλά εν περιπτώσει. Αφού γίνανε και σήμερα, έχει καλώς. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να κάνει το επάγγελμα που θέλει. Και η ικανοποίηση που αποφέρει αυτό είναι αναμφίβολο. Θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Δεν θα πρέπει παρά την κρίση να αποποιήσουμε την καλή ποιότητα ζωής την οποία θέλουμε να ζήσουμε. Εγώ θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες, αλλά πιστεύω ότι αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι και η κατάρτιση των εκπαιδευτών, των εκπαιδευτικών. Μπορούμε πολλά να κάνουμε ακόμη. Και αν δεν μπορούν να είναι στο ύψος τους οι εκπαιδευτικοί θα έχουν προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν τα νέα μέσα, τα ηλεκτρονικά και της πληροφορικής να είναι προσβάσιμα σε όλους, και στους εκπαιδευόμενους και στους εκπαιδευτές. Το να μάθει, κανεί, το να μάθει κανείς πώς να μαθαίνει επίσης είναι σημαντικό και πολλές φορές και σήμερα είναι κάτι το οποίο αγνοούμε. Η διδακτική αν θέλετε είναι κάτι το οποίο δεν μαθαίνεται εύκολα στα παιδιά σήμερα. Υπάρχουν κάποιες διδακτικές, παιδαγωγικές μέθοδοι που σήμερα έχουν παραγνωριστεί. Αλλά δεν πρέπει αυτό να το παραγνωρίζουμε. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το θέμα επίσης της ευθύνης του καθενός κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής του στην κάθε κοινωνία θα πρέπει να το επισημάνουμε επίσης. Και βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν στα πλαίσια της συνεχούς κατάρτισης μία υποχρέωση για όλους. Διότι πρέπει να εξοικειωθεί κανείς με αυτή την ιδέα της εφόρου ζωής μάθησης. Μία τελευταία παρατήρηση. Πιστεύω ότι θα πρέπει στα πλαίσια της επαγγελματικής κατάρτισης να γίνουν προσπάθειες ώστε η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να γίνει ακόμη πιο εύκολα. Ο Χάνς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια για την εξαιρετική εκθέση γνωμοδότηση και όλες αυτές τις ε, σκέψεις που μας υπέβαλε. Μπορώ να την υποστηρίξω πλήρως και όπως είπε ο κύριος Τσβέρ πρόκειται για κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει 10 χρόνια πριν αλλά εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει. Το 2010 στα πλαίσια της στρατηγικής 2000 θα έπρεπε να είχε και η οικονομία της Ευρώπης προχωρήσει και οι τεχνολογίες των πληροφοριών το ίδιο. Πολλά μπλα μπλα, αλλά ελάχιστα αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν ίσως στην Ευρώπη να ξανασκεφτούμε όλα αυτά τα θέματα που άπτονται της παιδείας. Επίσης, ελπίζω ότι δεν θα κάνουμε μόνο μια ακαδημαϊκή θεωρητική συζήτηση, αλλά θα καταλήξουμε σε συγκεκριμένα διατάφτα. Πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με μεγάλη πρόκληση, λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα τα οποία διαθέτουμε. Εδώ ο ρόλος των κρατών μελών είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτά τα σχέδια ή τα προγράμματα. Η Κομισιό στην ε, ανακοίνωσή της αυτή για τον ε, επανασχεδιασμό της εκπαίδευσης φτάνει την κατάλληλη στιγμή, διότι βρισκόμαστε εν μέσω οικονομικής κρίσης, την οποία πρέπει να ξεπεράσουμε, πρέπει να επιβιώσουμε και γνωρίζουμε ότι μία από τις ουσιαστικές ιδέες για να ξεπεράσουμε την, κρίση είναι την κρίση να επικεντρωθούμε στην εκπαίδευση και στην καινοτομία. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας και να γίνουμε ισχυροί ανταγωνιστές σε σχέση με τις υπόλοιπες δυνάμεις του κόσμου. Είναι λοιπόν στρατηγική σημασία στο θέμα αυτό και το έγραφο της Κομισιό είναι ένα πολύ καλό για εργαλείο για τα επόμενα χρόνια. Το χαιρετίζω και πρέπει να πω ότι κατά πρώτο λόγο να εξεπλάγει θετικά με την έκθεση αυτή. Η εκπαίδευση, επαναλαμβάνω, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όπλο στα χέρια μας για την ανάπτυξη και την πρόοδο. Και όπως είπε και η Πρόεδρος, οι αρχές επί του προπολογισμού, παρόλο που το θεωρούν πολύ σημαντικό, δεν του δίδουν τα κατάλληλα χρόνια. Πολύ συχνά πρόκειται για ευσεβείς πόθους. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει τα λόγια να τα κάνουμε πράξη. Πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τον επανασχεδιασμό της εκπαίδευσης. Επαναλαμβάνω, όχι κενά περιεχομένου λόγια. Εγώ έχω πει πόσες φορές είναι σημαντική, πόσο πολύ είναι η σημαντική είναι η εκπαίδευση για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Κοιτάξτε μόνο ποιες είναι οι ανάγκες που υπάρχουν και θα μπορούσαμε στα πλαίσια της ανοιχτής συνεργασίας να προχωρήσουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε και την αξία της εκπαίδευσης και της παιδείας αφευτεί, Δηλαδή, όχι μόνο για να συντείνει στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά ευρύτερα. Και θα ήθελα η παιδεία επίσης να εξεταστεί και από πολιτιστικής πλευράς. Η εκπαίδευση των ενηλίκων επίσης είναι πολύ σημαντική και η εκπαίδευση των παιδιών για να γίνουν αύριο όριμοι και χρήσιμοι πολίτες στην κοινωνία στην οποία ζουν. Την κοινωνική πτυχή επίσης και διάσταση του όλου προβλήματος αυτός θα πρέπει να εξεταστεί. Να μην εστιαστούμε μόνο στο ε, στενό συσχετισμό εκπαίδευσης και αγοράς της εργασίας. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε καλύτερα από σήμερα να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές και να μάθουμε ημένα από τους δε. Όπως είπε και η συγγήτρια, οργάνωσε κάποιες συναντήσεις τρογγυλής τραπέζης και εγώ οργάνωσα μία τέτοιου είδους συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφορούσε την κατάρτιση των εκπαιδευτών. Είχαμε εκπροσώπους από τα κράτη-μέλη αλλά πρέπει να πω ότι όλοι βγάλανε ένα χαρτάκι, διάβασαν το μπλα μπλα μπλα τους. Είπαν όλοι ότι εδώ έχουμε καλύτερα συστήματα από τους άλλους, εδώ έχουμε το καλύτερο σύστημα. Δεν ήθελε κανένας να μάθει τίποτα από τον άλλο, αλλά να του διδάξει αυτά που ήξερε. Όλα αυτά δεν είναι και πάρα πολύ εποφελή. Ελπίζω λοιπόν ότι τώρα θα μπορέσουμε να μάθουμε ένα από τους δε, να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές και θα ήθελα και πάλι να, να καλέσω την εισηγήτρια σε ένα σεμινάριο υψηλού επίπεδου που οργανώνω στις 16 Μαΐου για την εκπαίδευση και τον επανασχεδιασμό της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Θα έχουμε πολλούς εμπειρογνώμενους που θα λάβουν τον λόγο και θα έχουμε και τον Υπουργό παιδείας της Ιρλανδίας. Βεβαίως και όλα τα άλλα μέλη της Επιτροπής είναι προσκεκλημένα. Προσβλέπουμε λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση για να συζητήσουμε περαιτέρω. Ε, Η Πέτρα, θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ θερμά την ε, Καταρίνα ε, για αυτή την, όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε και νομίζω όλα αυτά δείχνουν με απόλυτη σαφήνεια ότι όσον αφορά την παιδεία υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες. Οι ε, ιδέες υπάρχουν, ε, η εφαρμογή τους χωλαίνει. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια. Κονδύλια για να υπάρξει εφαρμογή τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στα κράτη-μέλη. Ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στα κράτη-μέλη. Παρ' αυτά πιστεύω ότι στην εκπαίδευση πρέπει να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις γιατί σε τελική ανάλυση το μόνο που κάνουμε είναι να πληρώνουμε εκ των υστέρων μέσα από τα συστήματα κοινωνική ασφάλισης. Εγώ πιστεύω ότι κάθε ευρώ που επενδύουμε στην εκπαίδευση μας εξοικονομεί πολλά άλλα χρήματα. Και αυτό είναι κάτι ε, το οποίο θα πρέπει να περάσει ως πολιτική στα κράτη-μέλη. Και βεβαίως ε, πολύ ωραία αυτά που λέει η Κομισιόν, υπάρχει κινητικότητα. Το κάνουμε αυτό, μόνο από την άλλη αφού η Κομισιόν μας παίρνει τα χρήματα που χρειαζόμαστε δημιουργείται πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ε, το κατά πόσον τα διαρθρωτικά ταμεία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερα γιατί αυτά τα κονδύλια είναι απολύτως απαραίτητα και στην επένδυση, στην παιδεία πρέπει να υπάρξει επένδυση. Εκεί ε, λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευτούμε καλύτερα ε, το τι υπάρχει. Πολύ, αυτά, πολύ καλά αυτά που είπες για την επαγγελματική κατάρτιση. Ίσως ε, ως πολιτικοί μπορούμε και εμείς μερικές φορές να συμβάλλουμε έτσι ώστε αυτή η φήμη ότι δήθεν η επαγγελματική κατάρτιση είναι χειρότερη από την πανεπιστημιακή, κατά πόσο αυτό ισχύει όχι. Ξέρω ότι αυτό συζητήθηκε ε, στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 είπαμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο η ε, επαγγελματική ή πανεπιστημιακή κατάρτιση και η τεχνική έχει την ίδια αξία όπως, όπως τα πανεπιστημιακά προγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό στα κράτη-μέλη να βοηθήσουμε έτσι ώστε να υπάρχουν ε, λογικά εκπαιδευτικά συστήματα οι επιχειρήσεις να συμμετέχουν, γιατί αυτές ε, είναι οι δυνάμεις που λείπουν. Και όλοι έχουν συμφέρον να υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις. Είμαι σίγουρη ότι το ίδιο σημαίνει και σε άλλα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν όλες αυτές οι καλές ιδέες ας ε, συμπεριληφθούν στην έκθεση έτσι ώστε να ελπίζουμε ότι τουλάχιστον ε, θα δώσουμε κάποια κίνητρα ε, στα κράτη-μέλη. Ίσως ε, στον τομέα αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα κονδύλια από ό,τι συνέβη μέχρι σήμερα. Και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό θα εξυπηρετήσουμε πολύ και τα συμφέροντα των κρατών μελών. Προέδρο, θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα από την πρακτική εφαρμογή. Εγώ ζω στα γαλλογερμανικά σύνορα ή γαλλο με συγχωρείτε, ή λουξεμβουργιανα ε, σύνορα. Και ο κομωτής μου μου είπε ότι κυρία Πακ δεν μπορώ, δεν μου επιτρέπουν να προσλάβω μαθητευόμενους Γάλλους. Γάλλους αποκλείεται μου είπανε. Γιατί θα πρέπει αυτοί οι μαθητευόμενοι να πληρώσουν φόρο όπως ακριβώς προβλέπεται στον κανονισμό, στους νόμους της Γαλλίας. Η Γαλλία όμως είναι στα πόδια μου. Ανοίγοντας ε, το μπαλκόνι μου βλέπω απέναντι τη Γαλλία. Οι νέοι λοιπόν ε, δεν έχουν ε, θέση στη Γαλλία, θα μπορούσαν να έχουν δουλειά σε εμά. Την Παρασκευή έχω κλείσει ένα ραντεβού με τους αρμόδιους και κάποια λίστα βρούμε. Τα κράτη-μέλη λοιπόν είναι εκείνα τα οποία συμπεριφέρονται εθνικιστικά. Και σας λέω, η πρακτική εφαρμογή λείπει. Μπορούμε να μιλάμε θαυμάσια για πολλά πράγματα, μόνο που η πρακτική εφαρμογή είναι μερικές φορές απαράδεκτη. Όταν μου είπε ο ιδιοκτήτης του κομμωτηρίου αυτά που μου είπε, του είπα μην τα λέτε και πολύ δυνατά γιατί θα απογοτευτούν όλοι για την Ευρώπη ή από το τι είναι η Ευρώπη. Παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ. Ε, κάπως δυσάρεστη πινελιά, θα προτιμούσα να ακούσω μία πιο αισιόδοξη παρέμβαση εκ μέρους σας. Βεβαίως θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Νεβεντάλοβα, δυσκολεύομαι να πω το όνομα, για τον ενθουσιασμό της κατά την προετοιμασία Ε, της έκθεσης. Ε, ήδη η Στρογγυλή Τράπεζα ε, είχε ως αποτέλεσμα να ακουστούν πολύ εμπλεκόμενοι φορείς. Αυτό είναι άλλωστε ο στόχος. Θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων φορέων, όλων των παικτών για κάποια ζητήματα και βεβαίως σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία στον τομέα αυτό. Βεβαίως ε, μας ικανοποιεί πάρα πολύ ε, το γεγονός ότι υπάρχει τόσο ε, θετική ανταπόκριση στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού της εκπαίδευσης. Για μας, ανασχεδιασμός εκπαίδευσης σημαίνει μία απόπειρα, όπως είπαν και κάποιοι συνάδελφοί σας εδώ στην Επιτροπή, είναι μία απόπειρα αύξησης της ευαισθητοποίησης σε άλλες σφαίρες της πολιτικής, ότι η εκπαίδευση έχει σημασία παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στον προπολογισμό. Αποτελεί μια προσπάθεια να μπει στο χάρτη της ανάπτυξης και της απασχόλησης η εκπαίδευση, ότι είναι σημαντικό για την απασχολησιμότητα και είναι γεγονός ότι... Ε, η εκπαίδευση έχει μια ευρύτερη αποστολή για την ενεργό συμμετοχή ε, του πολίτη, ε, όμως στο τρέχον πλαίσιο ε, έντονης ανεργίας ε, μεταξύ των νέων, πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να ασχολείται με το πώς η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορεί να προωθήσει την απασχολησιμότητα. Δεν ε, πιστεύουμε ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας, δεν θα το λύσουν η εκπαίδευση και η κατάρτιση, υπάρχει και η έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης που σταματά την Ευρώπη από το να έχει υψηλότερα ποσοστά απασχολησιμότητας. Όμως το ερώτημά μας είναι κατά πόσο διαδραματίζει το ρόλο που της αναλογεί η εκπαίδευση και η καρτάτρηση και γι' αυτό πιστεύουμε ότι σε κάποιους τομείς θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα πράγματα, θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις ε, με πιο προσωμιωμένο τρόπο. Εμείς πιστεύουμε ότι ε, συμπεριλαμβάνονται 7 τομείς προτεραιότητας ε, του οποίους ανέφερε, μεταξύ των οποίων τέλος πάντων αναφέρθηκε και η εισηγήτρια Υπάρχουν πρωτοβουλίες που θα ήθελε να χρησιμοποιήσει, να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να υποστηρίξει τα ε, κράτη-μέλη, γιατί εμείς ε, ως καταλήτες απλώς θα δράσουμε και θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις από τις δράσεις που έχουμε προτείνει. Η πρώτη δράση είναι να υπάρξουν μαθητείες, ε, εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω μιας νέας συμμαχίας ε, ε, για το θέμα αυτό, κάτι το οποίο θα δρομολογηθεί τον Ιούνιο στην, στην συνεδρίαση της Λιψίας. πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Έχουμε δει ότι υπάρχουν ορισμένα συστήματα ε, πάρα πολύ ε, αποτελεσματικά και τα κράτη-μέλη μερικές φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα στη συμμετοχή τέτοιου είδους, ε, σε τέτοιου είδους συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε μια άλλη πρωτοβουλία της Επιτροπής, παράλληλα με τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης, που είναι μια πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου για την εγγύηση για την νεότητα αυτό έχει άμεση σχέση βέβαια και με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το Συμβούλιο το συζήτησε προκειμένου να υπάρξουν συστάσεις του Συμβουλίου προς αυτή την κατεύθυνση. Συζητήθηκε στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ. Δεν ξέρω ακριβώς ε, πώς ε, γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει άμεση σχέση με τον ασχετισμό της εκπαίδευσης και της ε, συμμαχίας για τη μαθητεία. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να υποστηρίξουμε και να προωθήσουμε την ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Μία ακόμη δράση επερχόμενη είναι η χρήση της τεχνολογίας πληροφορίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ε, της τεχνολογίας ε, και των υπολογιστών, γιατί η τεχνολογία και η πρόσβαση στη γνώση είναι ε, δυνατή σχεδόν παντού όμως δεν λαμβάνει χώρα με τον τρόπο που θα επέτρεπε η τεχνολογία. Γι' αυτό θα θέλαμε να μπούμε σε μια συζήτηση με τα κρατη για το πώς μπορούμε να ε, το ε, ενθαρρύνουμε αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι οι τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνο την αριστεία και την ποιότητα, αλλά και βελτίωση της πρόσβασης, μεγαλύτερη πρόσβαση στην ε, εκπαίδευση και την κατάρτιση για χώρες που βρίσκονται περισσότερο στο περιεθώριο, ώστε να υπάρχει μια ισότητα στην εκπαίδευση εκπαίδευση και την κατάρτιση και τρίτη, μια τρίτη πτυχή το οποίο η οποία συνεχίζει τη δυσκολία κινητικότητας ε, διασυνοριακά που αναφέρατε κι εσείς, είναι μια πιθανή, ένα, μια, ε, ε, ένας ευ, πιθανός ευρωπαϊκός τομέας ε, δεξιοτήτων. Πάρα πολλά μέσα έχουν δρομολογηθεί για την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δύο παραδείγματα να σας δώσω. Το, πλαίσιο, το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων που το γνωρίζετε κι εσείς. Υπάρχει το, ε, υπάρχουν τα credit systems, υπάρχουν ε, ε, οι εγγυήσει ποιότητας στην ανώτερη και την ανώτατη εκπαίδευση. Αυτά τα μέσα συνειδητοποιούμε λόγω αυτής, αυτού του, της συγκυρίας του ιστορικού πλαισίου δρομολόγησής τους και οι περιφέρειες οι οποίες απευθύνονταν ε, έχουν ε, κάπως αποκλίνουν πλέον το ένα από το άλλο και ε, η διαπερατότητα μεταξύ των διαφόρων οδών δεν ισχύει πλέον και η κινητικότητα μεταξύ των σε διασυνοριακό επίπεδο δεν είναι απολύτως επιτυχημένη. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι να δούμε πώς τα μέσα που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να είναι πιο συνεπή και πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ τους. Ε, θα ακούσετε περισσότερα από μας ε, από, από στο μέλλον γιατί είναι κάτι το οποίο η Επίτροπος ε, θα ήθελε ιδιαίτερα να προωθήσει μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τα σχόλιά σας για τον ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης. Ευχαριστούμε που επικροτείτε τις αρχικές μας πρωτοβουλίες και ευχαρίστω να συνεργαστούμε περαιτέρω για να λάβουμε υπόψη με βεβαιότητα τις ανησυχίες και τις απόψεις Επιτροπής σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι είμαι ευγνώμων όλα αυτά τα χρόνια στην Κομισιόν που καταθέτει τόσες πολλές προτάσεις και που επίσης πέτυχε αυτό το πλαίσιο ποιότητας, γιατί χωρίς αυτό δεν θα ήταν καν δυνατόν να προχωρήσουμε στο θέμα της αναγνώρισης. Αλλά αν δει κανείς τις συνθήκες, αυτό δεν είναι δουλειά της Κομισιόν, δηλαδή η Κομισιόν ε, κάνει πράγματα που είναι σημαντικά και ευτυχώ το Συμβούλιο ακολουθεί. Αν όμως τώρα σκεφτώ ότι το Συμβούλιο είναι εκείνο που μίλησε για την εγγύηση για τους νέους, διαρωτώ με πού είναι η συνέχεια στον προϋπολογισμό. Επανερχόμεθα λοιπόν συνεχώς στο ίδιο θέμα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Κατερίνα, θες να μιλήσεις? Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ευχαριστώ για όλα αυτά που μου είπατε και μία παρατήρηση για τον κύριο Σβέρ ε, που δεν είναι βέβαια παρόν. Ε, θέλω να πω ότι υπάρχουν και πολλές άλλες πρωτοβουλίες που προτείνονται από το Κοινοβούλιο και ο επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να συνεργαστεί για να αποκτήσει τους εργαζόμενους που επιθυμεί. Εμείς λοιπόν θα στηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, πολύ ωραία. Κατερίνα, τον Ιούνιο θα έχουμε την έκθεσή σου και μετά το Σεπτέμβριο θα ψηφίσουμε. Το 14 τώρα Εχθές ε, στις συνεδρίες των συντονιστών συμφωνήσαμε για ορισμένα πράγματα και στα, τα στείλαμε με mail. Από ό,τι βλέπω συμφωνείτε. Στα διάφορα δεν υπάρχει τίποτα. Επόμενη συνεδρίαση στις 28 Μαΐου από τις 9 μέχρι τις 12.30 και το απόγευμα θα ξεκινήσουμε στις 3.30 ε, ε, λόγω της διάσκεψης των Πρόεδρων. Ευχαριστώ πολύ τους διερμηνείς, λέει για καλή όρεξη.